Señorías, del día tiene que ver el informe anual Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα για το επόμενο. Θα αρχίσουμε σήμερα το απόγευμα με την έκθεση του αγαπητού μου φίλου του κυρίου Τρεμόσα που θα μας μιλήσει, παρουσιάσει την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του 2010. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, συνέταξα ως μεσο φιλελεύθερος από τη Μεσόγειο την έκθεση αυτή. Πραγματικά είμαι δείγμα αυτής της τάξης. Πρέπει να σας πω ότι όσο φιλελεύθεροι και μεσογειακοί πιστεύουμε όλο και περισσότερο στο ευρώ. Εγώ πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι την άποψη και πολλών άλλων συναδέλφων που πιστεύουμε στο ευρώ. Και πρέπει να πω ότι θα είχε ιτηθεί πάρα πολύ στην πολιτική της Ισπανίας αν δεν είχε το ευρώ. This Η έκθεσή μου λοιπόν έχει ως εξής. Όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσεως, Χαιρετίζω την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Σχετική Τράπεζας στις αγορές του 2010 και τώρα το καλοκαίρι. Δεδομένου ότι είναι το πρώτο το και μοναδικό πιστοτικό ευρωπαϊκό όργανο που μπορεί να παρέμβει. Οι παρεμβάσει τη κατά την άποψή μου, διέσωσαν το ευρώ, διότι χωρίς αυτές η κατάσταση σήμερα θα ήταν χειρότερη, όπω είπε την προηγούμενη Δευτέρα ο κ. Λάγκεν. Επίσης εκφράζω στην έκθεσή μου τα όρια της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κέντρης Τράπεζας και πιστεύω ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να εγνοούμε ότι στον ισολογισμό της τράπεζας υπάρχει και μια μεγάλη έκθεση για τα ε, επικίνδυνα κεφάλαια. Η αντιμετώπιση της κρίσης από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικαιτέρως για τις χώρες που δεν έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις όπως η Ισπανία στην άποψή μας ήταν σωστή η παρέμβαση. Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, ξέρω ότι η φορολογική ε, πειθαρχία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ε, φορολογική ενσωμάτωση. Δεν πρόκειται να γίνει αύριο μια ανοιχτή. Κάθε χώρα θα πρέπει να αρχίσει να λύει το όλο θέμα, αλλά θα πρέπει να αρχίσει τη συζήτηση τώρα. Σημερίζομαι την άποψη του κυρίου Τχισέ και λέγω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας Ευρωπαίος Υπουργός ε, Οικονομικών για να συντονίσει φορολογική πολιτική και να χειρίζεται την αποδοτικότητα του ευρώ. Αυτή η κρίση που είναι κυρίως κρίση χρέους αποδεικνύει ότι στην νομισματική ένωση η φορολογική πολιτική και η δημοσιονομική πολιτική δεν, αφορά, δεν αφορούν μόνο τα κράτη-μέλη. Επίσης, τονίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Διάθεσης Κονδυλίων για να ανακουφίζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λέγω πόσο σημαντικός είναι σε Ευρωπαϊκός Οικονομικός Μηχανισμός. Είμαι υπέρ των ευρωομολόγων αν μπορούν να μειώσουν το κόστος του δανεισμού και συγχρόνως να επιβάλλουν κυρώσεις στο υπερβολικό δημόσιο χρέος κάθε ε, κρατών. Η συζήτηση για αυτά τα που αφορά περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ενωπήση έχει στενή σχέση με τις δραστηριότητες της τράπεζας και την, ε, επηρεάζει την αποτελεσματικότητά της. Αυτή η συζήτηση είναι κάτι το οποίο αυτή τη συζήτηση συζητείται από όλους, άρα θα πρέπει και εμείς το συζητήσουμε. Τελικά όσον αφορά τη διαφάνεια. Ζητώ τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Υπουργών Οικονομικών όπως γίνεται στην Αμερική, στη Σουηδία και στην Ιαπωνία. Θεωρώ ότι η, δημοσίευση των πρακτικών είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει. Δεδομένου ότι χρειάζεται να υπάρχει αξιοπιστία ευρωπαϊκή και για τα ε, κοινοτικά όργανα. Διότι έτσι μόνο θα μπορέσουν να γίνουν πιο αξιόπιστα και να τύχουν τη ε, υποστήριξη όλων των πολιτών. Η Νομισματική Ένωση λοιπόν δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της αν δεν έχουμε δημοσίευση των πρακτικών των όσων συζητώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν θα υπάρχει η υποστήριξη που χρειάζεται. Σας ευχαριστώ. Είμαι ανοιχτό στις ερωτήσεις, στα σχόλιά σας για να βελτιωθεί η έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ε, Σε ευχαριστούμε κύριε Τρεμόσα. Αυτή τη στιγμή, όχι, όντως, βλέπω κάποιον εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Μαν εκπροσωπεί τον κύριο Μίτσελ που είναι ο σχέδιος συζητητής, δεν είναι έτσι. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το ΕΛΚ πολύ ευχαρίστως λαμβάνει πάντα το λόγο. Τώρα, κατά πόσο ως Γερμανός μπορώ να ε, παρουσιάσω την άποψη της πολιτικής μου ομάδας, ε, δεν το γνωρίζω. Γιατί ειδικά για το θέμα της οικονομίας υπάρχει και, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στην ομάδα μας. Λοιπόν, εγώ ε, συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τη φιλελεύθερη άποψη του συναδέλφου μου. στη δική μου τη χώρα, παρά τις αντικσότητες, έχουμε μια καλή κυβέρνηση, η συνεργασία Γερμανών και φιλελευθερών έχει αποδώσει και μέχρι τις επόμενες εκλογές έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για να περιορίσουμε τη δυσπιστία που αναφέρεται κατά καιρούς Πολλοί λένε, μα τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Πιστεύω λοιπόν ότι το σημαντικότερο είναι να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία. Ε, το ότι παρενεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εγώ αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα σωστό, πολύ σωστό. Ο ε, πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γερμανία ε, σε έναν πανηγυρικό λόγο επισήμανε ότι ε, δεν μπορεί η Γερμανία να στηρίζει αυτή τη μόνιμη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εγώ έχω άλλη άποψη. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διορθώνει λάθη που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά πρέπει να ισχύσει και κάτι άλλο. Η ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να ε, δέχεται την κριτική, ακόμα και ναι, ανεξάρτητο θεσμό. Να λέμε ότι είναι ιερό και όσιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό είναι λάθο. Εμεί ω βουλευτέ ε, γι' αυτό υπάρχουμε, για να ασκούμε κριτική. Πιστεύω βέβαια ότι η ΕΚΤ έχει παρουσιάσει θαυμάσιο έργο και έχω κατά νου τι ταχύτατε παρεμβάσει το περασμένο όταν εκλήθη να παρέμβει. Το, τώρα για το ύψος αγοράς κρατικών ομολόγων, εκεί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όχι μόνο τη Δευτέρα, αλλά και σε πολλές άλλες ευκαιρίες. Ο κύριος ε, Τρισέ έχει επισημάνει ότι ε, δεν αγοράζονται μόνο κρατικά ομόλογα, αλλά υπάρχει και μέρημνα. Ε, μετά από αυτή την κίνηση να υπάρχει και εκταμίευση κονδυλίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που βρίσκω σημαντικό είναι όσον αφορά στο ερώτημα ποιοι θεσμοί ε, γίνονται υποδεκτοί και σε ποιου υπάρχει πρόβλημα, λέμε ότι η ΕΚΤ, ακόμα και αν ασκούμε κριτική, η ΕΚΤ λοιπόν είναι αυτό το καταπληκτικό ε, μόρφωμα το οποίο μας έχει κρατήσει όλους ενωμένους. Πολλές ε, κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως τοποθέτηση είχαν επανειλημμένα ευκαιρίες να αντιπαρατεθούν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά στη τελική ανάλυση ο πολίτη ωφελήθηκε. Και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Γι' αυτό λοιπόν η άποψη κύριε Σιγητά που έχει εκφραστεί επανειλημμένα ότι οι εκθέσει ε, ε, πρέπει να δημοσιεύονται, αυτό δεν το βρίσκω απόλυτα σωστό. Τώρα, το πότε θα αγοραστούν πια κρατικά ομόλογα ε, αυτό στη Γερμανία αφορά τον πρόεδρο της Bundesbank. Αλλά ε, η Γερμανία όπως ξέρετε και οι Ολλανδοί έχουν καταψηφίσει πολλές ε, αποφάσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι δημοσιογράφοι έτσι και αλλιώς είναι εκείνοι που δημιουργούν, δημιουργούν θόρυβο, προκαλούν θόρυβο. Ε, δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσον ε, αυτός ο δρόμος που προτείνεται είναι σωστός. Γιατί μέχρι τώρα αρνήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα. Εμείς ως ε, μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, στις συζητήσεις του Δεκεμβρίου ε, που γίνονται στη Φραγκφούρτη εκεί την τελευταία φορά μας είπαν ότι η ΕΚΤ δεν επιθυμεί να υπάρχουν παρεμβάσεις απ' έξω. Όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ είναι ένα συλλογικό σώμα και δεν πρέπει να εκφράζονται οι απόψεις του σώματος αυτού προς τα έξω σε γενικές γραμμές ε, θεωρώ ότι στην έκθεση αυτή καθίσταται απόλυτα σαφές ε, ότι όλοι συμφωνούμε πόσο σημαντική είναι η ΕΚΤ. Ε, προφανώς ε, θα πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών και μια Ευρωπαϊκή κυβέρνηση, αλλά πάντα υπό δημοκρατικό έλεγχο. Και εδώ παίζει ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι για να κάνει επίδειξη δυνάμεων, αλλά γιατί αυτό εξάλλου αναφέρει και η Λισαβόνα. Όπου υπάρχει κυβέρνηση, πρέπει να υπάρχει και έλεγχο και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο σωστό εταίρο. Συμπέρασμα λοιπόν, η προσέγγιση του συναδέλφου είναι σωστή φιλελεύθερη προσέγγιση και λίγο και χριστιανοδημοκρατική προσέγγιση. Τώρα οι άλλοι προφανώς θα θελήσουν να κάνουν τις δικές τους διορθώσεις στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή βάση συζήτησης και ως οικονομική πολιτική ως Οικονομική Επιτροπή ανέκαθεν πιστεύαμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί σωστά και οποτεδήποτε υπήρξαν διαφωνίες λύθηκαν εδώ με το διάλογο. Ε, κύριε ε, Ισηγητά, θα καταθέσω ε, κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά το οδηγό νήμα που διατρέχει την έκθεσή εγώ προσωπικά το εγκρίνω και θα σας στηρίξω, δεν μπορώ βέβαια να δεσμευτώ, για το σύνολο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαν. Και εγώ δεν ε, μπορώ να βρω κανένα πρόβλημα στην εξαιρετική έκθεση την οποία έκανε ο συνάδελφος από τη χώρα μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ω εισηγήτη Σκιώδη για τον, την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τρεμόζε για την πρόταση έκθεση. Κατόπιν τη συζήτηση που έγινε τη Δευτέρα με τον κύριο Τρισέ, νομίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση επιβεβαιώνει την σημασία την οποία έχει αυτή η έκθεση, ε, ακόμη περισσότερο γιατί ανατε... νιώθουμε ξανά τις αναταραχές στη ε, την Ευρωζώνη. Και πρέπει να δούμε τους ε, επαρκείς ε, μηχανισμούς για να βγούμε από την τρέχουσα κατάσταση, μηχανισμούς που πρέπει να εμπλέξουν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε μπροστά μας την αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όμως το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτός είναι ο πιο ε, σωστός τρόπος αλληλεγγύης και θεωρώ όπως και ο κύριος Τρεμόζα ότι η σημερινή κατάσταση μπορεί να σταθεροποιηθεί με την μεταβίβαση κάποιων μερών προς την Ευρώπη ε, ευρωομορολόγων που θα μειώσει το κόστος ε, των χρεών ε, με τον περιορισμό στα 60% του ΑΕΠ θα ενθαρρύνει έτσι την δημοσιονομική πειθαρχία. Συμφωνώ με την έκθεση σε ό,τι αφορά ε, την ανάγκη να έχουμε μια ενιαία ε, φορολογική πολιτική και ενός φορέα για την αξιολόγηση της πολιτικής ικανότητας. Μια κοινή στατική φορολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ένα εργαλείο το οποίο δεν θα ενθαρρύνει την κερδοσκοπία χωρίς να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα. Εγώ αναμένω μια επικοδομητική ε, συνεργασία με τον κύριο Τρεμόζα και με τους άλλους ε, συναδέλφους της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Κουτάσο, κύριος Έπιν ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Τρεμόσα για την σχέση έκθεση. Συμφωνούμε με το θέμα του phasing out των uh, περισσότερης διαφάνειας και της ε, μη εφαρμογής κάποιων μέτρων παραδοσιακής πολιτικής. Ξέρουμε ότι με τον τρόπο που ενεργεί η Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα αφιερώθηκε μόνο στην σταθερότητα των τιμών και έχει κατά κάποιο τρόπο υποσκάψει κάποιες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά παρενέβη ενεργά όταν άρχισε να αγοράζει τα ομόλογα από κάποιες χώρες μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέμεινε την, ε, ε, ίστατη ε, ίστατος οργανισμός στον οποίο θα μπορούσε να προσφύγει καθήκη και ξέρουμε όπως είπε και ο Γερμανός Υπουργός ότι υπάρχουν κάποιες αλήθειε αλήθειες σε αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Πράγμα το οποίο αρνήθηκαν κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί ελεύθερη δεν υπάρχει και συνοχή στην ίδια τη τράπεζα. Νομίζω όμως ότι οι παρατηρήσει του Γερμανού Προέδρου θα μας κάνουν σκεφτούμε κάποια πράγματα. Η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα ως Τράπεζα Εγγύσεων νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο υποσκάπιστη την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λεχθεί με σαφήνεια στέξη του Κοινοβουλίου. Ο ε, κύριος Τρισέ επίσης πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών για να εποπτεύει τις οικονομικές και νομισματικές πολιτικές και να μπορέσει να ε, ελέγχει και τον όλο νομισματικό ε, τομέα στην Ευρώπη και εκτός. Είπε ότι αυτό είναι μακροπρόθεσμο, δεν είναι για αύριο. Οι εκθέσεις, το σχέδιο έκθεσης που συζητούμε τώρα κατά συνέπεια, νομίζω ότι δεν είναι ακόμη όριμες αυτό είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει τον τρόπο με το οποίο ε, λειτουργούν τα ευρωπαϊκά όργανα. Προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό όργανο. Όλοι ελπίζουν ότι κάποια μέρα ε, Ήλπιζαν ότι κάποια μέρα ε, θα μιλήσει με μία φωνή η Ευρώπη, αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Τι θα γίνει με την ε, Κομισιό που θα την αφήσει πίσω ο Υπουργός Οικονομικών, αυτός ο Υπερυπουργός ε, Οικονομικών. Αυτό το οποίο μας λείπει δεν είναι ότι έχουμε έλλειψη υπουργών, αλλά έλλειψη εφαρμογή ε, των κανόνων που θεσπίζουμε. Και το ότι είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα ξεπεράσει το, το έλλειμμα μας, θα είναι κάτω του 3% των, των και αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν σεβάστηκε κανένας. Άρα το πρόβλημα με την νομοθεσία δεν είναι να την έχουμε, αλλά την εφαρμόζουμε σωστά. Επίσης πρέπει να δούμε ότι επανήλθε και πάλι, όπως όλο το καλοκαίρι, το θέμα της συζήτησης των ευρωομολόγων. Ο κύριος ε, Τραμός μας μίλησε για τους φιλελεύθερους Μεσογείου. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν και φιλελεύθεροι στη Βόρεια Ευρώπη. Άρα πρέπει να μιλούμε Ίσως για τους ε, φιλεύθερους του ελαιολάδου και αυτούς του βουτύρου. Εγώ μιλάω εκ μέρους των Γερμανών και των Ολλανδών που είναι κάθετα αντίθετοι προς τα ευρωομόλογα. Παρά το γεγονός ότι είναι ε, φιλελεύθεροι. Άρα ποιος είναι φιλελεύθερος εδώ μέσα να μου πει τελικά. Δεν υποστηρίζω τις ιδέες ε, που εκφράζονται υπέρ της ασφάλειας στα πλαίσια ε, και ε, τα ευρωομόλογα τα οποία θα μπορέσουν να είναι μια καλή εγγύηση για το έργο. Ίσως υπάρχουν περισσότεροι ε, κίνδυνοι και δημοκρατικής ανεξαρτησίας όταν κάποια χώρα πρέπει να εγγυηθεί τα, για τα χρέη κάποιας άλλης χώρας. Κάποιοι θέλουν ίσως να αποδυναθεί περισσότερο η Ευρώπη και ίσως πιστεύουν ότι δημιουργώντας περισσότερα χρέη στην Ευρώπη θα σωσεί η κατάσταση. Αν θέλει κάποια χώρα να εκδώσει ευρωμόλογα, στο κάνει. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία. Τους καλώ να εκδώσουν ευρωομόλογα. Καλή αρχή θα είναι αυτή. Αλλά δεν έχουν το δικαίωμα το θέμα αυτό να το επιβάλλουν σε χώρες μέλη που δεν τα θέλουν. Γενικά λοιπόν θα έλεγα ότι όχι στα ευρωομόλογα χωρίς να υπάρχει συνένεση από τα Εθνικά Κοινοβούλια ή δημοψήφισμα για νομιμοποιηθεί η συμμετοχή όλων των κρατών της Ευρωζώνης στο εγχείρημα αυτό της έκδοσης ευρωομολόγων. Ευχαριστώ. Ε, ε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πιν. Σίγουρα Δίδω το λόγο για μια εντελώ διαφορετική άποψη στον κύριο Γκίγκολ. Ε, Αφού άκουσα τις διάφορες παρεμβάσει και την εισαγωγή του Ραμόν Τερεμόσα που δεν μπορώ να πω ότι είμαι μεσογειακός φιλελεύθερος, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι μη σοβινιστής γερμανός πράσινος. Και πιστεύω ότι αυτή είναι ακριβώς μια στάση που είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη-μέλη που φαίνεται να δείχνουν καλύτερη εικόνα από οικονομικής άποψης ε, συγκριτικά στην Ευρώπη να λένε είμαστε κατά των ευρωομολόγων, είμαστε κατά αυτού, κατά του άλλου. Όμως εγώ πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι η κατάσταση είναι υπερβολικά σοβαρή για τόσο βραχυπρόθεσμη πολιτική. Ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το ευρώ, υπάρχει ένα σοβαρό συστημικό κίνδυνος στο σύστημα. Και σα ευχαριστώ που μιλήσατε ανοιχτά γι' αυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σοβαροί συστημικοί κίνδυνοι στον ισολογισμό της ΕΚΤ. Και η ΕΚΤ αναγκάστηκε να ε, λάβει δράση για την έλλειψη βούλησης από πλευράς των κρατών μελών και των πολιτικών να επιλύσουν τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωζώνη. Ως εκ τούτου, είναι λάθος να επικρίνει κανείς αυτόν που προσπαθεί να διασώσει την ΕΚΤ, διότι αυτό που έκανε την δεδομένη στιγμή η ΕΚΤ είναι ότι ανέλαβε ρόλο διασώστη και η εντολή τους, η πρωταρχική, όχι η μόνη εντολή της, είναι η σταθερότητα των τιμών και του, του, του, νομίσματος. Και για να διασφαλίσει αυτή τη σταθερότητα αναγκάστηκε να πάρει μέτρα που δεν τα είχε επινοήσει στην αρχή, αλλά δεν απαγορευόντουσαν. Δηλαδή, όποιοι ισχυρίζονται ότι αυτό είναι κατά του νόμου, δεν βλέπει την πρωταρχική εντολή της ΕΚΤ και δεν την λαμβάνει σοβαρά υπόψη και ο πρόεδρος μας εδώ κάνει λάθος. Το ίδιο και ο συνάδελφος Έπιν. Συνεπώς θα πρέπει να προσθέσει κανείς ότι δεν αγόρασαν ομόλογα στην, στο πρωτογενή αγορά. Στη δευτερογενή αγορά τα αγόρασαν με έπτωση. Ακούω πολλά να λέγονται για τον κίνδυνο που είναι πραγματικός. Απ' την άλλη πλευρά όμως αν έχουν δίκιο οι οικονομολόγοι που λένε ότι στην περίπτωση της Ιταλίας και της Ισπανίας έχουμε ε, μία επιδείνωση της αγοράς, τότε η ΕΚΤ θα κάνει κέρδη αφού αγόρασε αυτά τα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά. Κανείς δεν αναφέρεται στις ευκαιρίες που προβάλλονται. Δεν λέω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να χαιρετήσουμε και να χειροκροτήσουμε. Δεν είμαστε ευτυχεί που αναγκάστηκε να αναλάβει αυτό το ρόλο η ΕΚΠΕ. Δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχεί γι' αυτό. Αλλά δεν πρέπει να επικρίνουμε εκείνου που ανέλαβαν την ευθύνη. Και επίση θα συμφωνούσα με τη βασική γραμμή του εισηγητή που λέει ότι επειδή βλέπουμε αυτούς τους κινδύνους, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για ένα πιο ομοσπονδιακό σύστημα στην Ευρωζώνη, ακριβώς γιατί θέλουμε να προστατέψουμε την έκτα από το να πρέπει να αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Θέλουμε και συμμερίζομαι αυτά που γράψατε, θα πρέπει να κινηθούμε προς ισχυρότερη ε, ενσωμάτωση της οικονομικής πολιτικής. Με όλα όσα αναφέρατε. Συμφωνώ με τον Τόμας Μαν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ε, με τον κοινοτικό τρόπο. Δεν μπορεί να το προσαρτήσουμε ε, με διακυβερνητικό τρόπο δίπλα στα ευρωπαϊκά όργανα. Το λέω και ως Γερμανός. Γιατί δεν είναι δυνατόν να εφευρίσκουμε νέες δομές από τις ε, γαλλογερμανικές συνόδους κορυφής. Θα πρέπει να αναπτυχθούν με βάση το σκεπτικό της κοινότητας. Και είμαι βέβαιος ότι ο εισηγητής έχει επίγνωση του θέματος και ο κύριος Έπινγκ έχει δίκιο. Ε, γνωρίζει ο εισηγητής ότι χρειάζονται να γίνουν αλλαγές στη συνθήκη και αυτό αληθεύει και ισχύει. Όμως ε, θα ήταν σωστό να πούμε ότι μετά από τα διδάγματα αυτής της κρίσης και του περιορισμού της διαχείρισης τη Ευρωζώνης μέσω συνόδων κορυφής πρέπει να δούμε τις σοβαρές επιπτώσεις και θα συμφωνούσα με τον εισηγήτη σε αυτό. Έχω κάποια θέματα ίσονος σημασίας για αριθμού. δεν θέλω να τα παραθέσω εδώ αναλυτικά, αλλά θα ήθελα να ε, αφού ε, ε, χαιρετίζω τα γενικά θέματα ορισμένα σημεία κριτικής. Πιστεύω ότι είναι αμφίβολο κατά πόσο η ΕΚΤ αναφέρθηκε στις τρεις ομάδες της Τρόικα να ήταν πάντα ο παίχτης ο οποίος όχι μόνο επέβαλε τη μεγαλύτερη πειθαρχία, ε, αληθεύει ότι οι χώρες που αυτή τη στιγμή ε, παίρνουν χρήματα από τον ε, μηχανισμό FSF που είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα θα πρέπει να επιδείξουν πειθαρχία. Αλλά και εκείνοι ήταν οι παίκτες που ήταν οι λιγότερο ευαίσθητοι στα κοινωνικά προβλήματα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να υπάρχει πειθαρχία αλλά ένας καλός φιλελεύθερος θα πρέπει να είναι και φιλελεύθερος θα πρέπει να γίνεται ίση κατανομή των προβλημάτων και ιδιαίτερα ε, από αυτούς που κέρδισαν πολλά πλούτη και πολλά ιδιωτικά πλούτη κερδίθηκαν και είναι χαρακτηριστικό. Τώρα στην Ιταλία πρέπει να το πούμε. Ένα μέτρο το οποίο καταργήθηκαν ήταν ε, ο φόρος ε, που δεν είδαμε ακριβώς στο, στο πρόγραμμα, δεν έγινε σωστή η κατανομή Πρέπει να προσθέσω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε θέματα όπως την εξωτερική αξία του ευρώ και τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της εξωτερικής αξίας. Χωρίς την ε, κρίση του ευρώ, πολλές εξωτερικές χώρες θα είχαν πολύ περισσότερα προβλήματα. Άρα υπάρχει και οικονομικός λόγος να επιφεληθούμε αυτού του πλεονεκτήματος κατακλείδη, θα έλεγα ότι στο θέμα της νομισματικής πολιτικής υπάρχουν προβλήματα στη δημιουργία ιδιωτικού χρέους. Το κείμενο δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Ε, σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, ε, είναι πολύ περισσότερο υπέρ του δημόσιου χρέους και ε, πρέπει να δούμε και το ιδιωτικό γιατί αναλήφθηκαν κινδύνοι μέσα από τις φούσκες ε, των επενδύσεων σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων και ε, μετά αναλήφθηκαν από το, το κράτος και οδήγησαν σε σοβαρά δημόσια χρέη. επειδή πολλές από τις χώρες που τώρα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα προϋπολογισμού δεν είχαν πρόβλημα προηγουμένως. Ας ε, κοιτάξουμε την Ισπανία και την Ιρλανδία. Αυτά οι χώρες είναι τα θύματα προβλημάτων στην αγορά των ιδιωτικών χρεών και μετά αντιμετώπισαν δυσκολίες και τώρα έχουν χρέο. Πολλέ χώρες είχαν καλές εξέλιξεις. Ακόμα και η Ιταλία μείωσε την έκθεσή της στο δημόσιο χρέος. Θα συντάξουμε κάποιες τροπολογίες για εμείς για τα νέα εργαλεία πολιτικής, της νομισματικής πολιτικής. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Η ΕΚΤ κοιτάει περισσότερο από τη δική μας προπτική ε, για το πληθωρισμό που δεν μπορεί να ελέγξει. Ε, ο συμπληθωρισμός ήταν μόνο στο 1% τον περασμένο χρόνο, για παράδειγμα. Με την νομισματική πολιτική δεν μπορείς να σταματήσεις τις ε, επιπτώσεις της ανόδου των τιμών των τροφίμων και των πόρων. Από την άλλη πλευρά, η ΕΚΤ δεν κάνει μεγάλη ανάλυση για τον πληθωρισμό των τιμών των περιουσιακών ε, στοιχείων. Στην αντιμετώπιση της κρίσης χρειάζεται, χρειάζονται χαμηλά επιτόκια, όμως δεν θέλουμε να έχουμε και φούσκες ε, ακινήτων. Και θα πρέπει να σκεφτεί πιο καινοτόμες μεθόδους. Θα σταματήσω εδώ και θα συντάξουμε περισσότερες τροπολογίες. Προσβλέπω στην ανταλλαγή απόψεων αλλά για τα βασικά ευρωπαϊκά ζητήματα έχω ακούσει να υπάρχει συμφωνία για την κοινοτική μέθοδο, την ανάγκη για περισσότερη ε, ε, συνεργασία, ιδιαίτερα για την προστασία της ΕΚΤΑ αθέμητη κριτική και για την ανάληψη κινδύνων και η σωστή ανταπόκριση και αντίδραση εδώ δεν είναι να γίνεται αυτή η κριτική, αλλά να δούμε τις επιπτώσεις ε, ε, στην κατεύθυνση την οποία εισηγείται ο εισηγητής. Ναι. Λέω, διάβασα την έκθεση του συναδέλφου για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον προηγούμενο χρόνο. Έχει εύστοχες παρατηρήσεις και κάνει και ορισμένες προτάσεις που πρέπει να συζητηθούν. Όμως εμένα αγαπητοί συνάδελφοι εντύπωση μου έκανε η αιτιολογική έκθεση του συναδέλφου που γράφτηκε πρόσφατα με βάση τις εξελίξεις και αυτή η αγωνία που βγάζει κατά μία έννοια και στην προφορική παρουσίαση είπε είμαι Μεσόγειος, είμαι φιλελεύθερος αλλά η αγωνία του δεν ήταν ενός Μεσογείου και ενός φιλελευθέρου ήταν η αγωνία ότι ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι προβλήματα έχουν τα γνωστά pinks κατά πλειοψηφία χώρες της Μεσογείου, όχι όλες. Τώρα το πρόβλημα, όπως εμφανίστηκε, το έχει και η Ισπανία, το έχει και η Ιταλία. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για Μεσόγειο με την παλιά έννοια. Μιλάμε για μια γενικευμένη ευρωκρίση και από την άλλη πλευρά, αν μου επιτρέπετε, και το φιλελεύθερος και οι άλλοι πολιτικοί προσδιορισμοί ενδεχομένως δεν έχουν και τόσο μεγάλη αξία αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί σήμερα διότι η κρίση δεν έχει περάσει και διότι βρισκόμαστε μπροστά στο πρόβλημα της κατάρρευσης, κατά τη γνώμη μου, του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, το κουβεντιάσαμε προχθές. Ακούστε λοιπόν τώρα τη γνώμη ενός αριστερού, όπως θέλω να πιστεύω, Μεσόγειου, σχετικά με το θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά τη γνώμη μου, αγαπητοί συνάδελφοι, αποδείχθηκε ότι ο καταστατικός στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή η σταθερότητα των τιμών, αντικειμενικά και μπροστά στα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, είναι καταστροφικός. Είναι καταστροφικός. Όχι μόνο όπως αποδείχθηκε, πράγμα γνωστό κατά μία έννοια, δεν εξασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα ούτε και την νομισματική σταθερότητα. Επομένως τίθεται θέμα καταστατικών στόχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ένα, και δεύτερο, το λέει κατά μία έννοια ο συνάδελφος, κατά τη γνώμη μου απαιτείται και πολιτικός δημοκρατικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσο αφορά τη συγκυρία και το 2010, ενδεχομένως γιατί γίνεται μια συζήτηση, γράφει πολλά ο τύπος, με αφορμή και την προχτεσινή κουβέντα, θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έναντι των άλλων θεσμών της Ένωσης κράτησε ή κρατάει την καλύτερη ή και τη σταθερότερη στάση. Δεν θα ήθελα να το αξιολογήσω αυτό. Θέλω όμως να αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις ευθύνες για το διάστημα που συζητάμε και θέλω σύντομα να σας τις αναφέρω. Πρώτον, έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν έβαλε φρένο στην έκρηξη των σπρέντς των επιτοκίων σε μια σειρά χώρες και θα μπορούσε να το κάνει αυτό αγοράζοντας περισσότερα κρατικά ομόλογα εγκαίρως και μπορούσε να το κάνει αυτό χωρίς να αλλάξει ούτε καμιά συνθήκη, ούτε να γίνει καμιά διακυβερνητική διάσκεψη, αλλά επειδή ο πληθωρισμός ήταν χαμηλά, θα μπορούσε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθεωρήσει την απόφαση του 1998 για πληθωρισμό γύρω στο 2% να πει επειδή έχουμε κρίση το όριο ανεβαίνει και να αγοράσει περισσότερα ομόλογα. Το δεύτερο, και είναι σημαντική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν έβαλε φρένο στη μαφία των κερδοσκόπων και εννοώ μαφία των κερδοσκόπων με όλη την ευθύνη και το έχουμε ξανασυζητήσει, δηλαδή στους οίκους αξιολόγησης που συνεχώς παραβαίνουν κατά καταστροφικό τρόπο, εδώ το έχουμε ομολογήσει όλοι και όχι μόνο δεν έβαλε φρένο πέρασε και τη δράση τους και τις εκθέσεις τους μέσα στο καταστατικό της ενώ είχε επισημανθεί το πρόβλημα. τρίτο δεν προσπάθησε να βάλει φρένο στην επανεμφάνιση της ύφεση που ζούμε αυτή την περίοδο διότι κρατάει υψηλότερα των ηνωμένων πολιτειών και της μεγάλης βρετανίας το επιτόκιό της. και τέταρτο δεν έβαλε φρένο στην επικίνδυνη μεγένθηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος που τα σημάδια δείχνουν ότι ενδεχομένως να αποτελέσει τη νέα μεγαλύτερη ενδεχομένως κρίση, φούσκα, μετά τα κίνητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυρία Λαγκάρτ για άλλη μια φορά επιμένει ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η ρευστότητα στις τράπεζες. Ε, εδώ αναζητούνται λύσεις που θα κάνουν τις μικρότερες δυνατές ζημιές. Επομένως, για να μην ε, σας κουράζω περισσότερο, φυσικά θα τα πούμε και στην αναλυτική εξέταση, νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε αντικειμενικά και μπροστά στα προβλήματα που έχει η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τη δική μας άποψη θα, θα θέλαμε να υπογραμμιστούν ορισμένα ή αυτά τα σημεία που εν συντομία ήθελα να πω στην πρώτη τοποθέτησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χουντή. Θα ήθελα τώρα να λάβω το λόγο. Και μετά έχουν ζητήσει το λόγο και άλλοι τρεις συνάδελφοι. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να πω το εξή. Πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι διαπίστωση των συμβάντων. Και η διαπίστωση είναι ότι Τη στιγμή την οποία δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση και δημιουργήσαμε το ευρώ, είχαμε άλλες απόψεις. Μετά είδαμε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα. Η θεσμική αρχιτεκτονική, όπως είπα, βασίστηκε σε τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα, ε, συγκεντρωτική νομισματική πολιτική, που ανατέθηκε σε μία κεντρική τράπεζα ανεξάρτητη μέσω τη συμφωνίου συνοχής μίας ανεξαρτησίας και ανοιχτή μέθοδος που δεν προέβλεπε αυτή που δεν θα τηρούσαν τις αρχές να υποστούν ακυρώσεις. Αυτές είναι οι τρεις, αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι ε, κανόνες οι οποίοι ήταν κατά την άποψή μου σαν τις ε, τρεις αρχές που βρίσ, πίσω από τις οποίες βρισκόταν η πόρτα του κόλασης του Δάντη. Είχαμε όμως προβλήματα όπως η μερική στάση πληρωμών της Ελλάδας, άλλα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουν άλλες χώρες της Μεσογειακής Ευρώπης. Άρα είχαμε ε, μη τήρηση αυτής της ε, πειθαρχία οι οποίες είχαμε. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν να μπορέσουν οι χώρες οι οποίες ε, ε, δεν μπορούν ε, να πληρώσουν όλα τα κριτήρια, να υφίστανται την πειθαρχία την οποία τους επιβάλλουν χωρίς να είναι σε θέση να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σύμφωνα με την σύμβαση την οποία έχουμε ανταγωνιστικότητα ώστε να μπορέσουμε να ε, υλοποιήσουμε αυτά τα οποία είπε στην έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, θα πρέπει να επιτρέπουν στι χώρε αυτέ να ανακουφιστούν από το χρέο το οποίο έχουν. Κατά την άποψή μου, ελέγχθη ότι τα ευρωμόλογα και ελέγχθη αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει ε, στα, στους άσωτους ιούς οι οποίοι δεν θέλουν να πιστούν και να ακολουθήσουν τις αρχές κάτι να κάνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα του οδηγήσει να μην ε, υφίστανται τι πιέσει των πολύ υψηλών επιτοκίων που θέλουν να επιβάλλουν κάτι. Δεύτερον, όπω είπε και ο κύριο Τρεμό, θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιε προποθέσει για τι χώρε οι οποίε δεν μπορούν να φτάσουν στο όριο το οποίο προβλέπεται. Και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε, αν δεν υπάρχουν ε, οι δυνατότητες ε, να πειθαρχήσουν στις σχετικές αρχές κάποιες χώρες να ε, μην μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υποστούν κάποιες κοινώσεις. Τρίτον, ε, τα ομόλογα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ειδικούς λόγους και να, να υπάρξουν και κάποιες, κάποιοι κανόνες για τα κράτη τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιήσουν αυτά τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Δίδεται η εντύπωση ότι θα υπάρξουν κυρώσεις οι οποίες θα πλήξουν κυρίως ε, τα διάφορα ταμεία συνοχής, διαρθρωτικά και θα... Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πλήξει περισσότερο τις χώρες που αποφελούνται από αυτά τα ταμεία. Αυτό όμως είναι εντελώς παράλογο. Διότι είναι σαν να λέει ότι κάποιος ότι εάν έχουμε πρόβλημα θα κλέψουμε τους φτωχούς για να μπορέσουμε να πληρώσουμε. Ο κύριος, όπως είπε και ο κύριος ε, Τρεμόσα, θα πρέπει να έχουμε ε, μία κεντρική ε, οικονομική πολιτική, προσέχοντα τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει όλε τι εξουσίε στα χέρια του και να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η ΕΚΤ έχει δυνατότητε μεγάλε δανειοδότηση, στα δύο τρίτα όλη τη Ευρώπη. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες δαδισμού που δίνουν, χωρίς να πούμε σε υπερβολές. Εγώ ως Μεσόγειος λοιπόν και ως χριστιανδημοκράτες πρέπει να πω ότι συμφωνώ πολύ περισσότερο με τον εισηγητή παρά με αυτά τα οποία ε, έγιναν από κάποιους ε, συναδέλφοι ακόμη και από την δική μου πολιτική έννοια. Διότι όπως λέγεται πολύ σωστά, η βάρκα δεν πλέει αριστερά ή δεξιά, αλλά έχει κέντρο στη μέση και έτσι κανονίζει την πορεία της. Ευχαριστώ. Well, since... Κύριε Σκυλακάκης, επειδή όλοι μιλάνε ε, για τους φιλελεύθερους Μεσογείου, ε, και εγώ θα μιλήσω ως ένας εκπρόσωπος αυτού του σπάνιου είδους Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η αποτυχία στο οικοδόμημα του ευρώ οφείλεται σε δύο στοιχεία. Το ένα είναι βέβαια στη ισόρρευση του χρέους, του χρέους. Το σημαντικότερο όμως αίτιο είναι ότι υπάρχει διαφορά ε, στον, στο ρυθμό ποσοστό παραγωγικότητας ανάμεσα στο βορρά και τον νότο. Αυτά είναι τα βαθύτερα αίτια. Και γι' αυτό το λόγο οι αυτόματες κυρώσεις είναι κατ' ουσίαν η μόνη λύση για το οικοδόμημα του ευρώ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές διαφορές ως προς ε, το ρυθμό της ε, παραγωγικότητας ε, που θα υπάρχει διαφορά τα επόμενα δέκα χρόνια όπως υπήρχε και κατά τα τελευταία δέκα χρόνια Πρέπει να ζητηθούν και άλλοι τρόποι, όχι μόνο οι αυτόματες κυρώσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση του Ραμόν ε, είναι, αποτελεί μια πολύ καλή αρχή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ο αποπληθωρισμός ως ένας τρόπος αντιμετώπισης διαφορών παραγωγικότητας δεν είναι σωστός τρόπος. Είναι πολύ δύσκολο για τα πολιτικά συστήματα να εφαρμόσουν αποπληθωριστικά μέτρα σε μία χώρα. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί την ε, λύση εφαρμογής του ευρώ και τη λύση της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Το άλλο που θέλω να πω, το τρίτο. Οι διακυβερνητικές πολιτικές έχουν εγγενείς δυσκολίες. Υπάρχουν εκλογές στις χώρες μας και οποτεδήποτε υπάρχουν εκλογές οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να κερδίσουν αυτές τις εκλογές. Και διακυβερνητική συνεργασία σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για τις κυβερνήσεις ε, που πρέπει να ε, συμφωνηθούν, άρα δηλαδή υπάρχουν και πάρα πολλές δυνατότητες για να προκύψουν παραβιάσεις. Εδώ το ευρώ και η σχετική πολιτική ε, στηρίζεται πάρα πολύ σε διακυβερνητική συνεργασία. Ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει το πρόβλημα αυτό να το αντιμετωπίσουμε περισσότερο, ουσιαστικότερα. Ε, τώρα, δύο θέματα επί της εκθέσεως και θα πω και κάτι άλλο που αφορά σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως είναι η Ελλάδα. Δύο θέματα για την έκθεση. Αναφέρθηκε ο Ευρωπαίος Υπουργό Οικονομικών. Πολύ καλή ιδέα, εντυπωσιακό ο τίτλος ε, και στην πολιτική πάντα ε, χρειαζόμαστε λέξεις κλειδί που τραβάνε την προσοχή, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι στην πραγματικότητα οι αρμοδιότητες αυτού του Υπουργού θα μοιάζουν με τις αρμοδιότητες ενός Πρωθυπουργού. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερα στοιχεία για να κατανοήσουμε αυτό το μελλοντικό αξίωμα και να καταλάβουν και άλλοι τι ακριβώς εννοούμε. Ε, γιατί στην Ευρώπη δεν έχουμε Ευρωπαίο Πρωθυπουργό. Κατόπιν, όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς οίκους αξιολόγησης, επειδή λοιπόν υπάρχει ε, ολιγοπόλιο οίκων αξιολόγηση, αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Και αυτοί οι οίκοι ε, δεν έκαναν καλή δουλειά. Όμως, οίκος αξιολόγηση αν υπάρχει, μετά την αρχική ε, σύστασή του. Δεν μπορεί ο οίκος αυτός ε, να ε, συντηρείται από κρατικά κονδύλια. Αυτό θα είναι γελίο. Δηλαδή θα πληρώνουμε κάποιον για να, λένε, για να λέει στις αγορές τι καλά που τα πάνε οι κυβερνήσεις. Αν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, ο οίκος αυτός θα πρέπει να είναι σοβαρός, να πουλάει τις απόψεις στην αγορά και μόνο έτσι θα μπορεί να λειτουργεί. Και θα ήταν χρήσιμος ένας τέτοιος οίκος εξελόγησης γιατί σας είπα υπάρχει αυτό λιγοπόλιο των ήδη υφιστάμενων οίκων εξελόγησης που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και τέλος, πώς φτάσαμε εκεί. Άκουσα την παρέμβαση του πράσινου συναδέλφου για την ανάγκη αναδιανομής. Κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό σε όλες τις χώρες. Εντάξει, στην Ιρλανδία ή αν θέλετε στην Ισπανία ε, και είχαμε επενδυτικές φούσκες. Στην Ελλάδα όμως δεν ήταν το ίδιο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα προκλήθηκε από χορήγηση κονδυλίων, κρατικών κονδυλίων σε ανθρώπους που είχαν πρόσβαση σε αυτά. Βλέπετε λοιπόν ότι η κατάσταση ποικίλει, δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες. Ο κύριος Λαμπέρα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά αυτή την έκθεση, θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Αυτό που εμένα μου λυπεί ε, και θα ήθελα να υπάρχει είναι να υπάρχει άλλη μία παράγραφος, θα το πω, ε, χοντροκομμένα και μετά μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Κοιτάξτε, τη Δευτέρα που ήρθε ο Τρισέ είπε κατ' ουσίαν ότι οι αγορές, ε, ο διατραπεζικός τομέας ε, είναι πλέον δυσλειτουργικό γιατί λόγω του δημόσιου χρέου, και αν τακτοποιηθούν τα δημόσια νομικά, θα πάνε όλα καλά και εντωμεταξύ μέχρι να γίνει αυτό είπε ο, ο, ο Τρισέ ότι η προσφέρει ρευστότητα στην αγορά. Όταν το ρωτήσαμε ε, για το πώς μπορεί να γίνει αυτός ο χειρισμός ε, των χρεογράφων και της τιμής των ε, χρεογράφων, κατ' ουσία οι απαντήσεις που έδωσε ο Τρισέ και πάλι είναι ανύπαρκτες. Μέσα στην ΕΚΤΕ πιστεύουμε ότι υπάρχει μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Εγώ ε, διπλωματικά ε, θα έλεγα ότι αυτό ενισχύει την ε, δυνατότητα ανάλυσης της ΕΚΤ. Δεν έχω κατά νου το να χαλαρώσει η πειθαρχία, αλλά εγώ λέω πρέπει να εξετάσουμε θέματα που είναι λιγάκι πιο περίπλοκα. Αυτά που λέξαμε προηγουμένως για τα, για τα ιδιωτικά χρέη. Αυτά είναι ένα καλό παράδειγμα. Ε, Αναφέρεται ότι δεν είναι σημαντικό παράγον, ενώ ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Σε πολλέ χώρε τα ιδιωτικά χρέη είναι το 200% του ΑΕΠ και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάτι, μια σχετική παράγραφος για να βελτιωθεί η έκθεση. Εγώ ε, νιώθω περίεργα, εκεί στην παράγραφο 14 λέτε ότι η ΕΚΤ πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να βασίζεται στην αξιολόγηση των οίκων, σε εκτιμήσει των οίκων αξιολόγηση. Κοιτάξτε, κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο οι αποφάσεις της ΕΚΤ να συναρτώνται από εκτιμήσεις ιδιωτών. Για να το πω ειλικρινά, λαμβανωμένων υπόψη όλων αυτών που ελέγχθησαν, την ανάλυση της ΕΚΤ, εγώ την ε, πιστεύω καλύτερα από τις ε, εκτιμήσεις ε, των οίκων αξιολόγησης. Έτσι λοιπόν, οι αποφάσεις της ΕΚΤ να είναι συνάρτηση της εκτίμησης οίκων αξιολόγησης, αυτό δεν είναι καλό. νομίζω σε γενικές γραμμές ότι θα είχαμε καλύτερη συζήτηση για τους οίκους αξιολόγησης αν δεν τους επιτρέπαμε αυτόματα να παρεμβαίνουν και αυτοί στην, ε, στην ε, νομοθεσία, στο νομοθετικό έργο. Όταν ένα ας πούμε λέει ότι εδώ πρόκειται για σκουπίδια, κατ' ουσίαν λέμε σε όλους τους ε, παίκτε σε παγκόσμιο επίπεδο ότι αυτό που ε, αναφέρουν οι οίκοι αξιολόγηση σχετικά με τα σκουπίδια, αυτό συγκεκριμένα ξεχάστε το. Ο Γιάν, ο Έπινγκ λέει ότι ε, πρέπει να προσθέσουμε περισσότερου θεσμού. Κοίταξε, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επίπεδα θεσμών. Όταν όμω μιλάμε για τον Υπουργό Οικονομικών τη Ευρώπη, θα μπορούσε να είναι ο ε, Επίτροπος ε, του ΕΚΟΦΗΝ Εκείνο λοιπόν που είπε ο συνάδελφό μα ο κύριο ε, Σκυλακάκη, είπε ότι ο Υπουργό Οικονομικών δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει και πρωθυπουργό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όμως και ο κύριος Τόμασμάν είπε Πρωθυπουργό δεν μπορεί να υπάρχει χωρί ε, Κοινοβούλιο. Εξάλλου ο Υπουργό Οικονομικών απλά καταθέτει τον προπολογισμό και μετά το Κοινοβούλιο αποφασίζει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό παράγον. Επανέρχομαι στον Γιάν. Ε, εσύ λες ότι τα ευρωομόλογα θα οδηγήσουν σε ε, πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη και είπε ότι μερικοί το επιθυμούν αυτό και εμεί όχι. Ε, εγώ δεν νομίζω ότι το θέλω αυτό, αλλά το χρειάζομαι αυτό, το χρειαζόμαστε αν πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε από εμά, οποιαδήποτε χώρα, αν θέλουμε οποιαδήποτε χώρα ή πιστεύουμε ότι μπορεί να βγει αλόβητη από την κρίση, όποιος το πιστεύει αυτό πλανάτε πλάνιν ικτράν. Μέχρι την αρχή πιστεύαμε ότι η, Γερμανία ε, θα τα πήρε μια χαρά, όλοι οι άλλοι θα καταστρέφονται. Ε, μετά όμως είδαμε ότι και αυτό δεν λειτουργεί. Αν πιστεύετε ότι οι Φλαμανδοί θα τα καταφέρουν καλύτερα, κάνετε λάθος. Και επειδή η οικονομική μας μοίρα, η μοίρα όλων μας είναι άρκτες οι μοίρε συνδεμένες ε, μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου και στις Βρυξέλλες παραδείγματος χάρη ε, που δεν είναι τέλεια πόλη. Βρισκόμαστε εδώ γιατί τη χρειαζόμαστε, τη χρειαζόμαστε για να υπάρχει ε, κοινωνική ευημερία. Το θέμα το οποίο τίθεται είναι όχι τι θέλουμε, αλλά τι χρειαζόμαστε. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοι, είπα, βρίσκω και εγώ ότι είναι μια σωστή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας η έκδοση του συναδέλφου. Η τράπεζα καλή δουλειά έχει κάνει, αλλά βεβαίως υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να τονίσουμε. Είχαμε πει και λέμε και τώρα ότι η αξιολόγηση ε, των διαφόρων οίκων δεν είναι κάτι το πολύ απλό, δεδομένου ότι επηρεάζει όλο τον κόσμο. Επίσης, τι θα συμβεί τώρα. Με αυτά που συμβαίνουν θα αλλάξουν κάποιες αποφάσεις σε σχέση με ένα άλλο θέμα τώρα. Η πίεση της τράπεζας κατά της αναδιάρθρωσης. Ήταν κάποια στιγμή προφανές ότι οι τράπεζες έπρεπε να δείξουν ότι οι κυβερνήσεις έπρεπε κάτι να κάνουν για να επιλύσουν το πρόβλημά τους με επιτυχή τρόπο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κοινή κατανόηση εκ μέρους όλων τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, θα πρέπει να αναφερθούμε στην πρακτική που ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν κάποιες χώρες. Δηλαδή, να βάλουν ανώτερο όριο στο χρέος τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να, να το προσέξουμε ιδιαίτερος. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το ζητήσει όταν ελέγχει την κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ ε, σκληρό να γίνει. Και τι μπορεί να κάνει στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση τράπεζα όταν βάζουμε ανώτοτο όριο. Βεβαίως χρειαζόμαστε ένα φορολογικό όργανο, όργανο το οποίο θα εποπτεύει, θα ελέγχει το τι μπορούν να κάνουν, να μην κάνουν οι διάφορες χώρες μέλη. Αλλά το να τα καπελώσει κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά ε, μία, ε, ένα κεντρικό όργανο νομίζω ότι ίσως δεν είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πολύ καλή στα χαρτιά η τράπεζα, αλλά στην πράξη είναι Μία τράπεζα που προσπαθεί να σώσει το ευρώ. Άρα πολιτικοποιείται με αυτό το οποίο κάνει. Άκουσα τι είπε και ο κύριος Μαργκάλιο, άκουσα και αυτά τα οποία λέξαν για τις κυρώσεις, για τις εγκυρίες. Αυτά είναι ωραία αν τα συζητούσαμε πριν από πέντε χρόνια. Τώρα ξέρουμε ότι αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επινοήσουμε μια νέα αρχιτεκτονική για να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ όλοι Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ο Ραμόν είναι καλό φιλελεύθερο. Είναι προσθέμενη αξία του γεγονό ότι είναι πια από τη Βαρκελόνη, αλλά πάντα ήταν καλό φιλελεύθερο από αν προέρχεται. Νομίζω είναι βασικό για αυτέ τι χώρε τουλάχιστον τη δική μου, εκτό τη Ευρωζώνης, να μην οριστεί αυτή ω μια ευρωκρίση. Θα πρέπει να αναφερθεί ω κρίση του χρέου. Αλλιώ, κανεί δεν θα πιστεύει, τουλάχιστον στη χώρα μου, ότι το ευρώ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Και εγώ πάντα ήμουν πολύ αυστηρό στα δικά μου σχόλια στη χώρα μου. Η ευθύνη για αυτή την κρίση ε, να απόκειται στην κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Δεν είναι το ευρώ σαν σύστημα. Είναι οι μεμονωμένες κυβερνήσεις και δεν έχουν ε, εκπληρώσει τις υποσχέσεις τους. Και εάν ε, έχουμε αντίθετα επιχειρήματα, τότε έχουμε πραγματικά μεγάλο πρόβλημα στο να ε, διευρύνουμε το ευρώ. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω από το Ρώμα να με βοηθήσει, διότι αναφέρθηκε στα ευρωομόλογα συνεχώς. Έχει αναφερθεί τα τελευταία δύο χρόνια ως ένα σύμβολο της διάσωσης των πάντων. εγώ ψήφισα υπέρ του και προσπάθησα το καλοκαίρι να το μελετήσω. Μπορείς να μου δώσεις κάποια πιστικά επιχειρήματα για το λόγο για τον οποίο πρέπει να εισαχθούν τώρα αυτά αυτή τη στιγμή. Είναι ένα Μήπως είναι ένα σύμβολο ότι αυτό θα ε, επιλύσει τα τρέχοντα προβλήματα. Γιατί πρέπει αυτές οι χώρες που έχουν, αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα αυτή τη στιγμή, τη συντρέχουσα κατάσταση, γιατί θα πρέπει να συμπεριφέρονται ως αν το χρέος να κατανέμεται σε άλλες χώρες. Αυτό είναι το επιχείρημα που άκουσα ε, στη χώρα μου, αλλά όπως είπα, εγώ υπερψήφισα. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν λέμε ότι αυτός είναι ο, ο τρόπος διάσωσης της Ευρώπης. Ραμόν, εσύ στη σοφία σου ε, προσπάθησε να με πείσεις ε, για να μπορέσω κι εγώ να πείσω τους ανθρώπους ε, στη χώρα μου ότι δεν είναι ο τρόπος, τουλάχιστον δεν είναι ο μοναδικός τρόπος ε, να βγούμε από την κρίση. Σε ευχαριστώ όμως για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, και μια καλή έκθεση ενός φιλελευθέρου από τη Βαρκελόνη. Ευχαριστώ. Νομίζω ο λόγος σε εσένα, Ραμόν. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό γιατί ξέρω ότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και είναι φορτωμένα μέρες σήμερα το απόγευμα. Έχει φύγει ο κύριος Μπίνκα. Θα ήθελα να του πω ότι η Μεσόγειος δεν παράγει μόνο ελαιόλαδο. Μπορώ να του δώσω στατιστικές λέγοντας ότι η Μεσόγειος θάλασσα είναι τόσο σημαντική όσο και ο Ατλαντικός όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Και είναι και πάρα πολύ σημαντική για τις δυνατότητες που έχει η ναυσιπλοεία μας μεταξύ ε, Μεσογείου και ακτών της Αμερικής μεταξύ άλλων. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι η θέση μου είναι η προσωπική μου άποψη και δεν μπορώ εγώ να μιλήσω εξ ονόματος όλης ομάδας των φιλελευθέρων. Ξέρω ότι στην ομάδα μου υπάρχουν πολλά μέλη που ακολουθούν τη γραμμή αυτή, όπως ο πρόεδρος Βερχόφστατ, ο οποίος με συνεκτικό τρόπο τα δύο τελευταία χρόνια ζητά περισσότερη οικονομική ενσωμάτωση. Υπάρχουν όμως και άλλα μέλη που είναι πιο, έχουν περισσότερους ενδιασμούς, όπως ο Wolf Klintz, που ήταν εντελώς αντίθετος εδώ και έξι χρόνια και μου είπε πριν από δύο μέρες τι μελετώ αυτή τη δυνατότητα, εξελίσσομαι στην άποψή μου και ίσως καταλήξω και εγώ στα ίδια συμπεράσματα, αλλά είμαι ανοιχτός ούτως ή άλλως. Αυτό μου αρέσει από τις βόρειες χώρες. Η ανοιχτή τους ε, νοοτροπία. Να μάθουν, να γνωρίσουν καλύτερα και ενδεχομένω να αλλάξουν και άποψη. Ούτως ή άλλως. Ξέρω ότι μεταξύ των Γερμανών φιλελευθέρων υπάρχουν και κάποιες ευαισθησίες υπέρ του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Και ίσως ο φίλος μου, ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, θα συμμερίζεται περισσότερο από άλλους απόψεις μου. Τώρα, Υπάρχουν και άλλες θέσεις. Υπάρχουν και άλλα ομάδες που είναι υπέρ περισσότερης ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά υπάρχουν και άλλοι, ξέρω, που υποστηρίζουν τις απόψεις μου. Τώρα, η κρίση αυτή πρέπει να εκλειφθεί ως δυνατότητα να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή ενοποίηση και να εξυγχρονίσουμε τις λιγότερο αποδοτικές οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως στην περίπτωση της Ισπανίας. Αναμένουμε λοιπόν ηγεσία, ηγετικό ρόλο εκ μέρους της Γερμανίας, που είναι η ηγετική χώρα στην Ευρώπη για το θέμα αυτό, όπως είπε και ο Helmut Kohl που ήταν τρομερός ηγέτης τη Ευρώπης και ηγήθηκε του όλου εγχειρήματο του ευρώ. Περιμένουμε λοιπόν τέτοιε διαδικασίες να αναπτυχθούν. Δεν έχουμε χρόνο τώρα για να εξηγήσω κάποια πράγματα για τα ευρωομόλογα. Είπε ο, ο Λιρέν ότι αν εμείς θεσπίσουμε τα ευρωομόλογα η απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να έχουμε φορολογική πειθαρχία εκ μέρους όλων των κρατών μελών. Περιμένω λοιπόν να δούμε ποιο θα είναι το σχετικό κείμενο πρόταση Επιτροπής για το θέμα αυτό των ευρωομολόγων. Ευχαριστώ. Θεσμία κατάθεση τροπολογιών 8 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. 3 Οκτωβρίου εξέτασή τους ψηφοφορία τέλος Οκτωβρίου, στόχος για να ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα και τώρα προχωρούμε στην επόμενη έκθεση. Οι υποθήκες. Οι υποθήκες που αφορούν τα ιδιωτικά ακίνητα, συγγνώμη, τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως ιδιωτικές κατηγές. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι Ισπανός από τη Μεσόγειο, είμαι Ισπανός από την πλευρά του Ατλαντικού, λέει ο εισηγητής. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να συνδυάσουμε τα νερά όλων των θαλασσών, των ποταμών και των λιμνών γενικότερα. Οι συμφωνίες για, τα, για τις υποθήκες είναι το θέμα της εκθεσής μου. Αρχίζοντας θα πρέπει να πω ότι πρόκειται για έναν φάκελο, για ένα θέμα στο οποίο θα συμμετάσχουν και άλλες ε, επιτροπές νομικών υποθέσεων και προστασίας του καταναλωτού. Θα συνεργαστούμε άτυπα με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και έχω αναλάβει την ε, δέσμευση με τον ε, συντάκτη της Επιτροπής αυτής να συναντηθώ πριν να περάσουμε στις ψήφιση των τροπολογιών για να δούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία τους αφορούν εκείνους από την Νομική Επιτροπή περισσότερο και με τους συναδέλφους της Επιτροπής ε, Προστασίας του καταναλωτού θα έχουμε ενισχυμένη συνεργασία για το θέμα αυτό. Αυτό που κάναμε μέχρι τώρα είναι να δούμε ποιες είναι οι ζώνες αρμοδιότητας, οι αποκλειστικές κάθε επιτροπής και ποιες είναι οι κοινέ αρμοδιότητες που έχουμε. Βεβαίως, στην περίπτωση που έχουμε κοινέ αρμοδιότητες, τον ηγετικό ρόλο τον διαδραματίζει η δική μας Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Στην έκθεση που ψηφίστηκε του κύριου Πέρβης ε, σε συνεργασία με έκθεση με Δίνα το 2007 και μετά από την παρουσίαση ε, της ε, Πράσινης Βίβλου του 2005 για την ε, υποθήκες, το πιο σημαντικό θέμα εκ των υστέρων ήταν η Λευκή Βίβλος του 2007 εκ μέρους της Επιτροπής. Οι υποθήκες, όπως ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο ενισχύει την εσωτερική αγορά και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική. Η Λευκή Βίβλος παρουσιάστηκε όταν ε, ήδη είχε αρχίσει να εμφανίζεται η κρίση των subprimes της Αμερικής. Και τότε έγινε το λόγο για το θέμα της διαχείρισης του κινδύνου και για λογικό και σοβαρό τρόπο χορήγησης τέτοιου είδους ε, κονδυλίων για τις ε, υποθήκες και για σοβαρό δανεισμό. Όλες αυτές οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και αργότερα και εγώ ανανορίστηκα ως εισηγητής για το θέμα αυτό άρχισα να ασχολούμαι σοβαρά με το θέμα, κάνοντας σοβαρό διάλογο με τους ε, συναδέλφους των, ε, από τις άλλες ομάδες που έχουν οριστεί και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με όλους και τα μέλη της Επιτροπής μας. Είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να καταθεθεί για να βελτιωθεί η έκθεσή μου, για να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε ευρεία συνένεση και συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε στα πλαίσια της συναπόφασης σε συμφωνία με, το Συμβούλιο. Η έκθεση μου είναι αρκετά ε, γενική καταρχάς. Καναφέρω πρώτα απ' όλα πόσο σημαντική είναι η κατάσταση στην αγορά σήμερα και αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι εκατομμύρια πολίτες σήμερα επηρεάζονται από τις ε, υποθήκες σήμερα και από αυτού του είδους ε, τα κονδύλια τα οποία ε, δανείζονται. Δεδομένου ότι η ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντική στην Ευρώπη δεδομένου ότι όλα αυτά τα θέματα μπορούν και την ε, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την επηρεάσουν. Ξέρουμε ότι η εσωτερική αγορά είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένη και κυρίως το θέμα των ε, υποθηκών. Η συνεργασία διακρατική είναι πάρα πολύ περιορισμένη, άρα Πρέπει να πούμε ότι η αγορά παρά το γεγονός ότι είναι κατακερματισμένη συγχρόνως είναι και πάρα πολύ δίσκαμπτη στον τομέα αυτό και έτσι δημιουργούνται προβλήματα. Η τιμή της υποθήκης απ' την άλλη και αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό εξαρτάται από πολλούς, ε, το κόστος της χρηματοδότησης από την, τα επιτόκια, από τη, τα κέρδη των ε, επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον τομέα αυτό και θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να μειωθεί το κόστος της διαχείρισης και το διοικητικό κόστος δεδομένου ότι θα πρέπει πάντα όλα αυτά να γίνονται σταθμίζοντας πάντα τους κινδύνους που υπάρχουν. Και θα πρέπει, ξέρουμε ε, ότι κάθε κονδύλι να και, που δίδεται να επομίζεται και ένα κόστος. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει για να υπάρχει σωστή διαχείριση αυτού του είδους των πιστώσεων. Έχουμε την πρόταση της Επιτροπή, έχουμε δύο παραρτήματο, έχουν παρουσιαστεί πρέπει να πω πάρα πολλές ε, ε, ε τροπολογίες, σχεδόν 180 και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο πιο σημαντικό θέμα. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του χρέους. Η υποθήκη για τον καταναλωτή είναι ένα μέρος του χρέους αλλά όχι το πιο προβληματικό. Πρέπει να πω ότι οι καταναλωτές πολλές φορές είναι οι ιδιωτικοί, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τα λιγότερα προβλήματα από ό,τι οι επιχειρήσεις. Εγώ έστειλα μια επιστολή στον Επίτροπο λέγοντας του ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ σωστά τα θέματα του, ε, της πίστεως, τα θέματα της, ε, ε, των υποθηκών, χωρίς να ξεχνούμε κάποιες αρχές. Πιστεύω ότι στην παρούσα οδηγία τρία θέματα δεν έχουν εξεταστεί και με τις τροπολογίες μας πιστεύω ότι θα πρέπει να τα εισαγάγουμε. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με την ε, με τον ιδιωτικό τομέα και με την υπερχρέωση του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την κατανοητική πίστη. Διότι συνήθως μιλάμε για την υπερχρέωση του κράτους, για το δημόσιο χρέος, αλλά πολλές φορές ξεχνούμε το τι, κάνουν, τι συμβαίνει με τους ιδιώτες. Θα πρέπει όμως το ιδιωτικό χρέος των καταναλωτών να το εξετάσουμε και από μακροοικονομικής προβάσεις και από μικρο. Να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ποια είναι τα όρια που θα μπορέσουν να έχει και δεύτερον από διαρθρωτικής πλευράς θα πρέπει να δούμε το εξής. Είναι σωστή η χρησιμοποίηση της ε, υποθήκης. Η είπα και ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν να κάνουν κάποιες αλλαγές, αλλά εμείς θα πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε επίσης πώς αντιμετωπίζουν το όλο θέμα κάποιοι πιστοτικοί οργανισμοί οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορούσαν και οι ίδιες να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν θέματα τα οποία ακόμη δεν έχουν απαντηθεί στην έκθεση της, στην πρόταση της Επιτροπής. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι στην έκθεση αυτή υπάρχουν τρία κεφάλαια τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση Επιτροπής και τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να εξεταστούν τώρα. Ένα θέμα είναι ποιος είναι ο ρυθμός με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα και ένα άλλο είναι ποιοι είναι οι κατάλληλοι δρόμοι. Πρώτα απ' όλα, για να κάνει κανείς υπεύθυνη χορήγηση και λήψη λαντίων θα πρέπει να έχει την κατάλληλη παιδεία κατά κάποιο τρόπο βάσει σωστής ενημέρωσης που θα βασίζεται σε τρία στοιχεία. Σωστή ενημέρωση, σωστή παιδεία, οικονομική και τρίτον δυνατότητα ε, να υπάρχει κάποιος επαγγελματίας που να συμβουλεύει αυτούς οι οποίοι ε, θα πάρουν αυτό το δάνειο. Όταν μιλώ για παιδεία οικονομική αναφέρομαι σε γνώση του όλου θέματος εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Δεν μιλάω γενικότερα για ακαδημαϊκά. Δεύτερον, η πρόταση της Επιτροπής ασχολείται κυρίως με θέματα που οδηγούν στη σύναψη της σύμβασης για την χορήγηση της υποθήκης. Μπορούν εδώ να υπάρξουν βελτιώσεις αλλά όσον αφορά την αποπληρωμή του χρέους για τον ιδιώτη, δεν είναι σαφείς οι κανόνες. Άρα, υπάρχουν θέματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στους παρόντες κανόνες που ισχύουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο κεφάλαιο για την σωστή εκτέλεση όλων αυτών των συμβάσεων ε, που αφορούν την, ε, τις υποθήκες. Όχι μόνο για την ε, καταβολή ενωμέρους τους χρέους για την υποθήκη, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν κάποιοι κοινοί κανόνες. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι υπάρχουν στη Λευκή Βίβλο, άλλοι στην Πράσινη Βίβλο, και δεν υπάρχει ε, ενιαία, ενιαίο σύνολο κανόνων. Επίσης, τι γίνεται όταν κάποιος έχει μια υποθήκη για μια ιδιωτική κατοικία στη χώρα του, σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μετακομίζει. Υπάρχουν χιλιάδες θέματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως και η χορήγηση μιας ε, κάποιας ευελιξίας εκ μέρους των ε, τραπεζών που κάνουν αυτού του είδους τα δάνεια στους ιδιώτες. Ευελιξία για το σύστημα καταβολής των χρεών, δεδομένου ότι ε, δεν έχουν, ε, όλοι όσοι παίρνουν ένα τέτοιο είδους ε, νυπόθηκο δάνειο δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή δεν έχουν εισοδήματα κάθε τέλος του μηνός, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία έχω θέσει στην εκθεσή μου. Επίσης μίλησα για την ανάγκη να υπάρχουν μηχανισμοί για να διευθετούν το θέμα της χορήγησης ε, μιας υποθήκης σε ένα νόμισμα και να λαμβάνεται υπόψη μετά ισοτιμία αν πρέπει να πληρωθεί σε άλλο νόμισμα, ευρώ, μη ευρώ, φερρυπίν. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνονται μέσα σε ένα σύνολο κανόνων ώστε να μην υπάρχουν ε, ε, έκτακτα προβλήματα. Επίσης, τι γίνεται με την πρόορη εξόφληση κάποιου ενυπόθηκου δανείου, τι γίνεται σε περίπτωση οικονομικής κρίσης, ε, τι θα γίνει με όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Για όλα αυτά τα θέματα που αναφέρω θα πρέπει ε, να έχουμε σωστούς κανόνες. Επίσης, τι γίνεται με το θέμα της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αν θέλουμε το ευρωπαϊκό σύστημα να δουλέψει, θα πρέπει η χρηματοδότηση των υποθηκών και το θέμα των κεφαλαίων που διατίθενται να γίνονται μέσα στα πλαίσια ενός αξιόπιστου και διαφανού συστήματος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός ανιχνευσιμότητας και αξιολόγησης ώστε οι υποθήκες και τα ενυπόθηκα δάνεια να γίνονται με συνεκτικές μεθόδους και με διαφανείς μεθόδους για να λειτουργήσει σωστά η αγορά. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία περαιτέρω, ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όλο σύστημα χορήγησης ενυπόθηκων δανείων στην Ευρώπη. Επίσης, ξέρουμε ότι να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ε, ε, μηχανισμού όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη προς την αγορά. Στην πρότασή μου Επίσης αναφέρουμε στο θέμα του κινδύνου. Η πρόταση της Επιτροπής κατά την άποψή μου είναι σωστή, αλλά θέτει το πρόβλημα με κάπως ε, ομοιόμορφο τρόπο υπερβολικά. Εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα διάφορα τα ενυπόθηκα δάνεια έχουν διαφορετικού βαθμού κίνδυνο. Μπορούν να υπάρξουν ε, μεγάλες αυξομοιώσεις στον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι πιστώσεις για τα δάνεια αυτά. Άρα, ανάλογα με την αγορά στην οποία αναπτύσσονται, μπορούν να έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο ρίσκο. Los mercados. Identificar cuáles son los créditos hipotecarios que plantean mayores riesgos. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα και ένα σωστό οπλοστάσιο μέτρων που θα μπορούν να εφαρμόσουν ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που μπορούν να δημιουργηθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θα θέλαμε ενισχυμένες ε, αρμόδιες αρχές ε, ε, εποπτείας. Καλή είναι η εποπτεία και ο έλεγχος για θέματα πρακτικά και εγώ είπα ότι θα πρέπει να υπάρχει και ενίσχυση των αρχών στις οποίες βρίσκεται το αγαθό το οποίο έχει αποτελέσει το αντικείμενο του ενυποθήκου δανείου. Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες και δανειζόμενοι δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις αγορές τις οποίες βρίσκονται τα δάνεια. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία παρουσίασα στους συναδέλφους. Επίσης, πρέπει να υπάρχει μία περίοδος ε, χρόνου που πρέπει να δίδεται σε αυτόν ο οποίος υπογράφει το δάνειο να ενημερωθεί σωστά πριν να, είναι, ε, να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Θα πρέπει ο δανειολήπτης να είναι σωστά ενημερωμένος και να έχει τον κατάλληλο χρόνο να σκεφτεί και να μελετήσει αυτά που του προτείνουν για να μην χρειάζεται βάζοντα την τσίφρα του την επομένη το πρωί να αναλάβει δέσμευση. Θα πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Διότι είναι καλή όχι μόνο για τον καταναλωτή, αλλά και για την ίδια την βιομηχανία του κλάδου. Δεδομένου ότι κανένα μετά εκ των υστέρων δεν θα μπορεί να πει ότι αγνοούσε του κανόνε και δεν μπορεί να τιμήσει τι υποχρεώσει του. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρου κάποιον η κατάλληλη συμβουλή, επαγγελματική συμβουλή, ώστε που να δίδεται από επαγγελματίε δεδομένου ότι πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι κανόνες για τη χρηματοδότηση ώστε να μην ε, ε, δίδονται συμβουλές μόνο και μόνο για λόγους marketing. Αυτά είναι τα θέματα που ήθελα να σας αναφέρω. Θα επανέλθω γιατί σήμερα έχω πάρει πολύ από το χρόνο σας και θα ακούσω και τους ε, συναδέλφους και μετά θα επανέλθω. Τελειώνοντας την παρέμβασή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου για να κάνω την εκδεσή μου κυρίως τους δύο βοηθούς μου και την γραμματεία της Επιτροπής για την εξαιρετική βοήθεια που μου παρήχαν. Ευχαριστώ. Έχουμε πέντε ε, σκιωδησίγητες, έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας, πέντε συγητές και άλλους πέντε που έχουν ειστεί το λόγο. Εκτός από τους συγητές έχουμε... Και ο κύριος Νίτρας προστίθεται επίσης και θα κλείσω τον κατάλογο. Αν λοιπόν ε, κάποιος ε, άλλος θέλει να λάβει το λόγο, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν θα μπορέσει. Και ίσως οι, οι μπορούν να περιστούν σε τέσσερα λεπτά ο καθένας ε, και αν τηρηθεί αυτό θα τα καταφέρουμε να μιλήσουν όλοι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα σταματήσω και ένα λεπτό νωρίτερα και έτσι θα τηρήσω νομίζω το χρόνο. Κοιτάξτε, εγώ διάβασα την έκθεση και διάβασα και τις ε, τροπολογίες ε, που κατέθεσε ο συνάδελφος ε, Σάντσετς και παρουσιάζει το πρόβλημα κυρίως για, από το πρίσμα του πολίτη που θέλει να αποκτήσει μια υποθήκη. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιες σωστές λύσεις, θα τις όλοι. Εγώ συμφωνώ ότι ο πολίτης τη στιγμή που ζητάει ενυπόθηκο δάνειο ε, θέλει να έχει τις καλύτερες ε, δυνατές προϋποθέσεις, διαφάνεια κυρίως ε, στις διαδικασίες. Πρέπει όμως να αποφύγουμε και τις υπερβολικές ρυθμίσεις σε αυτό τον τομέα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Γιατί με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο άκαμπτη η αγορά και είναι πολύ πιο δύσκολο να χορηγηθούν τα δάνεια. Διότι η σχέση ανάμεσα στον κατασκευαστικό τομέα και τα ενυπόθηκα δάνεια είναι μια ξεκάθαρη ε, σχέση, οριζόντια θέση. Είναι η θέση, η σχέση ανάμεσα στην τράπεζα και τον πολίτη. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερες ρυθμίσεις, να αποφύγουμε όμως τις υπερβολικές ρυθμίσεις και την εισαγωγή αυτόματων κριτηρίων, τα οποία θα οδηγούσαν στο αντίθετο από το ευκταίο αποτέλεσμα. Οφείλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να είναι και πάρα πολύ συνετή. Να έχει κατά νου ότι θα πρέπει να προστατευτεί κυρίως ο πολίτης. Αυτά μάλιστα σε μια χρονική στιγμή όπως αυτή που διανύουμε τώρα. Ε, κατά την άποψή μας στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη ε, και ένα ε, τραπεζικό σύστημα το οποίο θα συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση. Το να το καταστήσουμε άκαμπτο, αυτό θα οδηγήσει στο να μπλοκάρουμε το σύστημα. Πρέπει να αποφευθούν οι πρακτικές εκείνες ε, οι οποίες οδήγησαν σε υπερβολικές ε, ρυθμίσεις, να αποφευθούν όλα εκείνα τα οποία παρουσιάστηκαν κατά προηγούμενα έτη. Η κρίση των ε, ενυπόθηκων δανείων δεν έπληξε την Ευρώπη. Ξέσπασε στι Ηνωμένε Πολιτείε και οι επιπτώσει ε, έγιναν στην Ευρώπη, αλλά ο τομέας όμως εδώ στην Ευρώπη διασώθηκε. Κατόπιν τούτου σίγουρα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση, όμως εκείνο που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να προστατευτεί ο καταναλωτής, να προστατευτεί η κοινή αγορά, να εφαρμάζονται ομοιογενείς διατάξεις και συναλφεστάνσεις. Αυτό πρέπει να αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα ε, κατασκευαστικών εταιριών που δεν οφείλονται στην ποιότητα και στο κόστος. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο. Το τρίτο που θέλω να πω ε, που κατά την άποψή μου και αυτό έχει άμεση σχέση με την ευρωπαϊκή κληρονομιά. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να διαφυλάξουμε ε, την αγορά των μικρομεσαίων επιχείρησεων και αυτό δεν θα το πετύχουμε με το να καθιστούμε άκαμπτη, όπως σας είπα, αυτή την ισορροπία που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο. Το δικαίωμα του καταναλωτή ε, να μπορεί να προεξοφλεί το δάνειο, επ' αυτού συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ λοιπόν ότι ε, θα πρέπει πράγματι ε, να ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν για την ε, έγκαιρη και προώρη εξόφληση δανείων. Το πρόβλημα είναι βέβαια οι τράπεζες, κατά πόσον οι τράπεζες συμφωνούν με αυτό. Τώρα, όσον αφορά το ότι θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να, να αποφασίζει μόνο του το τι θα κάνει το δάνειο, αυτό αφορά τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στην 102 και όλες οι υπόλοιπε. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Αναφέρομαι και στο ότι η επιχείρηση θα πρέπει επίσης ε, να έχει την ελευθερία να ε, διαπραγματεύεται το δάνειό της οι σχέσεις λοιπόν ανάμεσα στα, στις τράπεζες και τους πελάτες, αυτά είναι δύο τελείως διαφορετικοί Θα ήθελα όμως κλείνοντας να σε παρακαλέσω να μιλήσεις για τις ε, τροπολογίες, την 95, την 94 και την 96. Είναι τροπολογίες που αφορούν στην ε, προσφορά και πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε προσεκτικά την 152, 153, 157 σχετικά με την σύνεση που πρέπει να επικρατεί. Εκείνο λοιπόν που ενδιαφέρει είναι να εξετάσουμε τη σχετική οδηγία η οποία είναι απαραίτητη για να αποφεύγουμε επικαλύψεις. Θεωρώ λοιπόν, τελειώντας ε, κυρία Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, διαφορές, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Και σας λέω, εκείνο που ενδιαφέρει είναι τα ε, συμφέροντα του καταναλωτή, αλλά και των ελεύθερων επιχειρήσεων. Πρόεδρος, Ξέρω ότι όταν έχουμε μία τόσο μακρά ε, εισήγηση είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί κανείς σε λίγα μονολεπτά. Επόμενος εκ μέρους των Φιλιππέων ο κύριος Στάρξ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία. Πιστεύω ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι η αγορά των υποθηκών δεν ήταν ο λόγος πίσω από την κρίση του χρέους, αλλά ε, στις περισσότερες χώρες δεν είχαμε πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι με καλή προσέγγιση να πούμε ότι θα πρέπει να συντάξουμε μια έκθεση, αλλά θα έχουμε υπόψη αυτό που είπε ο Επίτροπος είναι ένα προκαταπτικό πρώτο στάδιο και το επόμενο στάδιο θα το λάβουμε αργότερα όταν θα δούμε τις περαιτέρω πτυχές. Ε, οι Επίτροπες θα έχει τα ε, περαιτέρω στάδια στο μέλλον να παρουσιάσει. Νομίζω ότι ο εισηγητής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ιχνηλασιμότητα, διαφήμιση κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και ο συντονιστικός ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη είναι πολύ καλή προσέγγιση. Έχω κάποια σχόλια. Ε, ο Παραλαλής σας είχε δίκιο όταν είπε ότι δεν πρέπει να υπερρυθμίζουμε. Όταν δούμε την ε, αξία και τα έσοδα, πόσο από αυτά τα έσοδα θα πρέπει να καταβάλλονται στην ε, εξόφληση του της υποθήκης. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε περιορισμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές αγορές, στο γεγονός ότι δεν τηρούνται ε, οι συνήθειες. Οι ε, τεράπεζες έχουν την ευελιξία στη διάθεσή του. Θα πρέπει να είμαστε σαφεί όταν ε, μιλάμε για υπερβολικά αυστηρά όρια. Θα πρέπει να αφήσουμε την αγορά να κάνει τη δουλειά της. Θα πρέπει να δούμε την, ε, στο πλαίσιο αυτό η ε, τροπολογία 75 αναφέρεται στην στα κράτη-μέλη που εξασφαλίζουν ε, η πολιτική θα πρέπει να είναι τους ίδιους του εργοδότες. Μπορεί εμείς να θέσουμε την αρχή, αλλά δεν πρέπει να πάμε παραπέρα, διότι αυτό μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά. Όταν μιλάμε για την διαφήμιση και λέμε όταν ένα οίκο αξιολόγηση κάνει μια διαφήμιση στο ραδιόφωνο, θα πρέπει να περιλάβει και κάτι και online. Δεν μιλάμε μόνο για διαφημίσεις σε, εντύπω υλικό. Θα πρέπει να έχουμε πλήρη παροχή πληροφόρησης. Εδώ όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες. Μπορεί να είναι να, έχουμε και συνδεδεμένες πωλήσει. Αν μιλάμε για ε, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί με μια υποθήκη, σημαίνει ότι μπορεί να έχει καλύτερους όρους είτε για το συμβόλαιο είτε για την υποθήκη. Ιδιαίτερα αν μιλάμε για τον ασφαλιστή ή αυτόν που παρέχει την πίστοση ή τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει σύνδεση ανάμεσα σε αυτά, αλλά δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Θα πρέπει όμως να είναι δυνατόν και αυτό θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Θα πρέπει να δώσουμε ευελιξία, όπως είπα και πριν. Αν λέμε ότι παρέχουμε ένα δάνειο, τότε κάποιος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και μπορεί να έχει μείωση του εισοδήματό του. Αλλά μιλάμε για ένα νέο άτομο στην αρχή της σταδιοδρομίας του. Το εισόδημα του μπορεί να αυξηθεί. Δεν αναφέρεται κάτι γι' αυτό στην τροπολογία 121 θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό και να ε, βεβαιωθούμε ότι είμαστε ευέλικτοι σε όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο σε τομείς που μπορεί να προκύψουν προβλήματα, αλλά και εκεί που μπορούν να δούμε ευκαιρίες για τους νέους. Έχω καλύψει ένα-δυο σημεία μέχρι στιγμής. Προσβλέπω στην συζήτηση και τη συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Φόρτ. Ευχαριστώ. Επειδή αυτό, αυτή είναι η μοναδική πιο σημαντική οικονομική απόφαση θα πρέπει εμείς ως πολίτες να λάβουμε, νομίζω θα πρέπει να έχουμε σωστά επιχειρήματα και λυπάμαι αν θα ξεπεράσει τα τέσσερα λεπτά, διότι είναι σημαντικό. Ευχαριστώ τον εισηγητή που ε, αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο σε αυτό. Και ειδικά που έχουμε δει το θέμα της οικονομικής εκπαίδευσης, πολύ σημαντικό και ε, επίσης τη διαφήμιση που να είναι αναλογική προς τα μέσα. Το θέμα για τις ε, ε, αρχές δικέ αρχές και εποπτείας που γνωρίζει καλύτερα την αγορά. Αυτό είναι σημαντικό θα πρέπει κάποιο να συμμορφώνεται με κανόνες και πρότυπα που είναι κατάλληλα στην δεδομένη αγορά. Ε, όπως είπε και ο προηγούμενο μιλητή, στο θέμα της πιστοληπτικής ικανότητας, της φερενκιότητας, αυτή, αυτή είναι η καρδιά της οδηγία. Τι, είναι ένα, ε, ε, ε, σε ποιον είναι σωστό να, να, να γίνει ένα δάνειο. Στο 121 πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν αποκλείονται κάποιες ομάδες, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι άτομα που μπορεί να έχουν εποχιακές επιχειρήσεις, μια ταβέρνα ε, ή κάποιος που έχει φάρμα μεγαλοπούλες. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ευελιξία ε, στους ε, ελεύθερους επαγγελματίους αυτοαπασχολούμενους με υπεύθυνο τρόπο. Ας δούμε την τροπολογία 121 και την πιστοληπτική ικανότητα γιατί είναι σημαντικό. Στην προπόληση και τις περιόδους προπόλησης είναι σημαντικό διότι για μια εταιρεία να κάνει μια ε, προσφορά ε, χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν σταθερή αποδοχή διότι οι τιμές της αγοράς ε, στις οποίες διακυμαίνονται θα πρέπει να έχουν μια σταθερή προσφορά που μετά γίνεται αποδεκτή για 14 ε, μέρες, τότε μπορεί να αυξηθεί η τιμή αυτής της προσφοράς. Αυτή η αβεβαιότητα, ιδιαίτερα σε χώρες όπου μπορεί να υπάρχουν αλυσίδες ε, πωλήσεων ή πληστηριασμούς, ε, που γίνονται προσφορές, διαγωνισμοί, θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Η, η περίοδος των 14 ημερών δεν είμαι πεπισμένη ότι αυτό έχει τεθεί σωστά στο κείμενο. Θα πρέπει να το δούμε ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει προ πληροφόρηση. Δηλαδή, ένας χρόνος όπου γίνεται, η προσφορά, γίνεται αποδεκτή η προσφορά και αυτό γνωστοποιείται. Στην αποκάλυψη πληροφοριών θα μπορούμε να το επεξεργαστούμε καλύτερα εδώ αυτό το σημείο, διότι υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο να δίνουμε πληροφορίες στους καταναλωτές, αλλά να μην τους υπερφορτώνουμε με πληροφορίες, διότι αν υπερφορτώνει τον καταναλωτή με πληροφορίες, τότε δεν βλέπουν την ουσία. Είναι σημαντικό να το δούμε και αυτό. Το, για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τι δικαιώμα έχω στην υποθήκη. Έχω. Ο εισηγητή έχει υποβάλει τι ε, από την 138 στην 144, από το δικαίωμα προπληρωμής, δικαίωμα να πάρω την υποθήκη όταν μετακομίζω, ε, δικαίωμα μεταβι, ε, μεταφοράς ε, μερικοί θέλουν αυτά τα δικαιώματα, άλλοι μπορεί να μην τα θέλουν. Αυτά τα δικαιώματα είναι δαπανηρά για αυτούς που παρέχουν τα δικαιώματα. Θα πρέπει να ε, βεβαιωθούμε ότι έχουμε ισορροπία κόστους αποτελεσματικότητας. Να μην είναι αναγκασμένοι όλοι να πληρώνουν για ε, μια υποθέκη η οποία περιλαμβάνει τα πάντα. Μ' αρέσει η έννοια του EMKI, του Ευρωπαϊκού Κωδικού Ενυπόθηκου Δανείου, του κωδικού. Είναι καλή ιδέα. Οι εταιρείε θα πρέπει να κρατούν αρχεία ε, σχετικά με το δάνειο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που προέκυψε σε διάφορα κράτη-μέλη. Όμως κάποια κράτη-μέλη ήδη έχουν πολύ αποτελεσματικά ε, ε, προγράμματα. δεν πρέπει να γίνει επικάλυψη σε κάποιες χώρες που ήδη υπάρχει, διότι αυτό επίσης εμπεριέχει επιπρόσθετο κόστος. Στο θέμα των προληπτικών διατάξεων 152 ε, είναι σημαντικά μέτρα, αλλά είναι πολύ χοντροκομμένα, όπως ε, για τους δείχτες δανείου προς αξία, χρέος προς περιουσιακά στοιχεία. Θα πρέπει στο 150, τροπολογία 150, να δούμε τις ιδιαιτερότητες ε, της κάθε αγοράς ακινήτων, των κάθε ακινήτων, των περιστάσεων του κάθε δανειζομένου. Αυτά τα μέτρα αποκλείουν ορισμένες, ορισμένα ακίνητα ή κάποιους δανειζόμενους. Στην διασταυρωτή πώληση κάποιων ε, προϊόντων βλέπω τι προσπαθείτε να πετύχετε εδώ αλλά ίσως να υπάρχουν και άλλοι τρόποι που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Στην 145 είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό, διότι δεν θέλουμε κάποιος να, ε, ε, ε, να βρεθεί έξω από το σπίτι του χωρίς λόγο. θα πρέπει να υπάρχει τρόπος διαπραγμάτευσης μιας κατάστασης ατόμων που έχουν οικονομικές δυσχέρειες στην εξόφληση του δανείου, αλλά με ανησυχεί το τέλος της παραγράφου όπου ε, υπονοείται ότι εναπόκειται στον τραπεζίτη να ορίσει τι σημαίνει επαρκές βιωτικό επίπεδο. Ε, δεν ε, μ' αρέσει αυτή η ιδέα του να ορίζεται αυτό το επίπεδο από τους τραπεζίτες. Θα πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση για αυτό το θέμα. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο Σβέν από τους Πράσινους. Συμφωνώ και εγώ ότι εδώ χρειάζεται σοβαρή και εντελεχής δουλειά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους μίλησαν ε, και τον εισηγητή για την έκθεση που αποτελεί μια πολύ καλή βάση για συζήτηση. Λόγω του ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, δεν θέλω να μπω σε όλες τις ε, λεπτομέρειες. Όμως, επιθυμώ να επισημάνω ορισμένα βασικά στοιχεία. Για μας, λοιπόν, η κρίση του ευρώ και η κρίση χρέους, όσον αφορά αυτά τα δύο στοιχεία, η σχέση ανάμεσα στην ε, αγορά πίστης ε, για ε, σπίτια αφενός και η μακροοικονομική σταθερότητα, η σχέση ανάμεσα στα δύο είναι καθοριστική σημασίας. δεν μπορούμε λοιπόν να παρακολουθούμε αυτήν την αγορά με τον ίδιο τρόπο όπως το κάναμε πριν από την κρίση, διότι εντωμεταξύ σε πάρα πολλά κράτη-μέλη, σε διάφορα κράτη-μέλη, ε, κρίση αυτή προκάλεσε σημαντικά προβλήματα. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Ρόγκοφ για την ε, χρηματοπιστωτική κρίση θα διαπιστώσετε ότι η αγορά ακινήτων και τα προβλήματα στις τράπεζες αυτοί είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην χρηματοπιστωτική κρίση. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν πάνω σε ένα θέμα. Οποτεδήποτε σκεπτόμεθα όλα αυτά, να μην ξεχνάμε τις μακροοικονομικές συνέπειες και πώς μπορούμε να επιφέρουμε στην έκθεση τη μακροοικονομική σταθερότητα. Από ό,τι άκουσα, η Κομισιόν δεν είναι πρόθυμη να περάσει πέρα από την να προχωρήσει πέρα από την εμβέλεια της έκθεσης που είναι η προστασία του καταναλωτή. Καλό, αλλά δεν αρκεί αυτό. Έχουμε πολλούς ε, μεγάλο εργολάβους ε, που συνέβαλαν και αυτοί στο να υπάρξει η φούσκα στην αγορά. Αυτοί όμως δεν αναφέρονται πουθενά και δεν προβλέπονται ε, αποτελεσματικά μέτρα για ε, αντικυκλικές ε, ρυθμίσεις. Ο συγητής με την 152, την 153, την 154 τροπολογία κάνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση όμως με αυτά που είναι απαραίτητα. Αυτά δεν αρκούν και γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε ποιο μέτρο ενδείκνυται περισσότερο απ' όλα για να επιτύχουμε την αντικυκλικότητα. Κατά τα άλλα βλέπουμε να υπάρχουν πολλές ε, καλές προτάσεις από τον εισηγητή που ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση κυρίως εκεί που γίνεται λόγος ε, για την ε, αποζημίωση οποτεδήποτε προσφέρονται δάνεια και κυρίως εκεί που γίνεται λόγος για την ενημέρωση του καταναλωτή. Αναφέρονται πολλά και σημαντικά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας την ε, ε, παροχή δανείων σε ξένο συνάλλαγμα. Αν διαβάσετε ε, την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι το κύριο μέλημά της σε πολλές σχόλες της Ανατολικής Ευρώπης. Να απασχολεί πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν ας ενημερώσουμε σχετικά και τους καταναλωτές. Πρέπει να σας πω ότι είμαι λιγάκι επιφυλακτικός όσον αφορά την δυνατότητα της πρόορης εξόφλησης. Εγώ είμαι ε, πιο κοντά σε αυτό που προτείνει η Κομισιόν, ότι η πρόορη εξόφληση μπορεί σε κάποιες αγορές κατοικίας να πρόκειται ακόμα πιο βραχυπρόθεσμες ε, πολιτικές στέγασης. Βλέπουμε όμως ότι η κυκλικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κατόπιν τούτου η πρόορη εξόφληση πρέπει να αντιμετωπιστεί κάτω από δύο πρίσματα. Αφενός τα δικαιώματα του καταναλωτή, αφετέρου όμως και η μακροοικονομική σταθερότητα. Αν ανοίξουμε διάπλατα την πόρτα στην πρόορη εξόφληση, ε, τότε θα έχουμε ε, μεγαλύτερη βεντάλια επιτοκίων και λιγότερη σταθερότητα στην αγορά. Εγώ λοιπόν είμαι επιφυλακτικός και θέλω το θέμα αυτό να το συζητήσουμε σοβαρά. Κατά τα άλλα, ε, θέλω να πω ότι προσβλέπω στην ε, καλή συνεργασία επί του θέματος. Ας προσπαθήσουμε το θέμα να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Θα ήθελα επίσης να ακούσω και την άποψη ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν ε, ο εισηγητής μπορούσε να ζητήσει την άποψη και αυτή τη Επιτροπή. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ ότι η προσπάθεια που κάνει ο εισηγητής και τον ευχαριστώ πολύ είναι και σοβαρή, είναι σε θετική κατεύθυνση. Επικροτώ και τις ενέργειες τις οποίες έχει κάνει και με τα περισσότερα από τα μέτρα που προτείνει, δεν θα τα αναφέρω για λόγους χρόνου, ε, συμφωνώ. Θα περιοριστώ σε μια γενική επισήμαση και σε δύο επιμέρους παρατηρήσεις, λιγότερο από τα τέσσερα λεπτά που δικαιούται ο καθένας μας, ε, διότι είναι σύντομος χρόνος. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι όποιες ρυθμίσεις και αν γίνουν, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν καλείται η αγορά να λύσει πάγιες και κοινωνικές ανάγκες με κερδοσκοπικά κριτήρια, τα αποτελέσματα θα είναι προβληματικά έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι ο πυρήνας του προβλήματος είναι η υπερδιόγκωση του ενυπόθηκου δανεισμού και η άμεση σύνδεση με τα καινοτόμα προϊόντα. Και εδώ, σε σχέση με τα καινοτόμα προϊόντα που δημιούργησαν και τη φούσκα και ούτω καθεξής, εδώ είναι το προβληματικό της όλης υπόθεσης και προφανώς δεν έχω την απέτηση η έκθεση να το αντιμετωπίζει αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και αυτό το θέμα δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να μας ξεφεύγει. Δύο επιμέρους παρατηρήσεις για αυτήν καθ' αυτήν την έκθεση. Ε, συμφωνώ είναι θετικά τα μέτρα. Υπάρχουν δύο κενά θα έλεγε κανεί που πρέπει να δοθεί απάντηση. Το ένα σημείο είναι ότι τι θα γίνει, υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους, ότι αφού το πρόβλημα δεν ήταν η αδυναμία των καταναλωτών να αποπληρώσουν τα χρέη και η ανεύθυνη δανειοληψία, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που έχουν συνεισφέρει, που έχουν συμβάλει στο πρόβλημα που υπάρχουν κενά και η έκθεση του συναδέλφου που Δηλαδή, τι θα γίνει με τις κατασκευαστικές εταιρείες, τι θα γίνει με τους οργανισμούς, τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις. Και το δεύτερο, ένα κρίσιμο κατά τη γνώμη μου θέμα, είναι αυτό των μεσιτών των πιστώσεων, μεσίτες πιστώσεων. Έχοντας υπόψη ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ε, με τους ε, καταναλωτές και που έπαιξαν και καταλητικό ρόλο στις ΗΠΑ. Η Επιτροπή από ό,τι βλέπω τους θεσμοθετεί και απλώς αν διάβασα καλά θεωρεί ότι είναι επαρκές να τους εντάξει σε ένα μητρό για καλύτερο έλεγχο. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι εκεί και δεν είναι μόνο εκεί και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Επομένω, θα χρειαστεί να δούμε και από αυτή την άποψη και στο σημείο αυτό τι πρέπει να γίνει. Περιορίζομαι σε αυτά γιατί ο χρόνο είναι περιορισμένο. Συμφωνώ όμω ότι είναι μια θετική προσπάθεια και ευχαριστώ και πάλι τον συνάδελφο. Uh, um, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τώρα άλλους έξι που έχουν ζητήσει το λόγο και τελικά αν χρειαστούμε πολύ χρόνο θα αναγκαστούμε τη συζήτηση να την συνεχίσουμε μετά την ψηφοφορία. Μπαστός θα δούμε τι θα κάνουμε. Η Αιλίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι πρέπει το θέμα να συζητηθεί περισσότερο. Ε, γιατί πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο τεχνικής φύσεως ε, τεχνικό θέμα. Μερικοί έθιξαν πολλά και σημαντικά θέματα. Εγώ θα περιοριστώ σε λίγα μόνο σημεία. Πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ λιγάκι όσον αφορά το ύφος της ε, συζήτησης. Υπάρχει περιττός σκεπτικισμός για το κατά πόσο πρέπει να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση στον τομέα ή όχι. Οι φιλελεύθεροι λένε ότι αυτό δεν είναι καλό για τον για την τομέα, για τις τράπεζες, αλλά θέλω να τους πω ότι αν δεν έχουμε ανταγωνισμό δεν θα προσφέρουμε τη δυνατότητα επιλογής στον καταναλωτή ε, και ο ανταγωνισμός είναι εκείνο που βοηθάει ε, και στον τομέα των πιστώσεων και των δανείων. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε την αγορά, να προσφέρουμε στον καταναλωτή ε, περισσότερες επιλογές. Επίσης πιστεύω Ξέρω, ας πούμε, η συνάδελφο Κάθριν Στήλα ε, δουλεύει πάνω στο θέμα. Ε, ξέρετε, στον τομέα αυτό ασχοληθήκαμε με κάτι παρεμφερές. Όταν είχαμε την οδηγία ε, περί πιστώσεων, χορήγησης πιστώσεων. Και τότε μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε τη βιομηχανία, αλλά μπορέσαμε και να προσφέρουμε και προστασία στον καταναλωτή. Δεν νομίζω ότι ε, πρέπει να γνωρούμε μερικά προβλήματα που πολύ σωστά ετέθησαν. Και εγώ χαιρετίζω το γεγονός ότι ο εισηγητής μπαίνει σε λεπτομέρειες, από ό,τι φαίνεται έχει διαβουλευτεί με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η εκπαίδευση είναι καθοριστική σημασία, πράγματι για να ξέρουν οι ε, καταναλωτές τι υπογράφουν. Ε, επιπλέον το θέμα της συγκρισιμότητας και αυτό είναι ε, πολύ σημαντικό είναι δυνατόν να καθορίσουμε γενικές αρχές, να γίνονται αυτές αποδεκτές και από τις, τους κατανοητές και από τη βιομηχανία. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά χρειαζόμαστε και κάποιες ε, στάνταρτ αρχές. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, τη μόνη περαιτέρω λεπτομέρεια που θέλω να φέρω είναι ότι στον τομέα αυτό έχουμε ενώσεις οι οποίες ε, παρέχουν ε, συμβουλές ε, και αυτές μάλιστα μερικές φορές χορηγούν και ίδιες επιστώσεις. Δεν πρέπει λοιπόν αυτές να αποκλείονται από την αγορά γιατί ίσως να υπάρχουν οι κανόνες που να τις οδηγήσουν έξω από την αγορά. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι τελικά πιστεύω πράγματι να επιτύχουμε ένα πολύ ικανοποιητικό νομοθέτημα. Ο Μάνουελ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να κάνουμε έκθεση πρώτα απ' όλα να κάνουμε κάτι που θα αρέσει και στην ε, Κομισιόν και στο Συμβούλιο και να το συζητήσουμε γρήγορα και δεύτερον να κάνουμε μια έκθεση που να προσθέσει μια κάποια να παρέχει μια κάποια προσθέμενη αξία όπως έγινε η έκθεση αυτή. Δηλαδή το να υπογραμμίσουμε κάποια θέματα ε, τα οποία είναι ε, θέματα όπως συγκεκριμένη περίπτωση που απασχολούν όλους τους ε, ε, καταναλωτές να μπορέσουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στην κατακαιρματισμένη χώρα να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το θέμα ε, του υπερβολικής υπεχρέωσης και τα θέματα της υπερβολικής έκθεσης όλων των πιστωτών σε όλους τους κινδύνους που δημιούργησε η οικονομική κίνδυση είναι κάτι το σημαντικό που κάναμε. Νομίζω ότι μπροστά, έχουμε, μπροστά μας έχουμε να κάνουμε με μία έκθεση που αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Άρα, διαφάνεια, σωστοί κανόνες και όλα αυτά τα οποία λέγονται στην έκθεση του συναδέλφου μου είναι σωτική σημασία. Είναι εξαιρετική σημασία η έκθεση και νομίζω ότι όλη η ομάδα μου την υποστηρίζει και θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι να ενεργούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για να παρέχουμε και να παράγουμε τη θέμενη αξία προτάσει Επιτροπή. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι έρχονται και άλλοι συνέλφοι στην αίθουσα για την ψηφοφορία. Ακόμη ένας ομιλητής λοιπόν και μετά θα πρέπει να αναβάλουμε για μετά την ψηφοφορία την ε, συνέχιση της συζήτησης. Ο το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος δεδομένου ότι δεν πρέπει να παρηγορούμε. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε συνεκτικότητα μεταξύ της νομοθεσίας για τις υποθήκες και της ε, των, καταναλωτικών, των ενυποθήκων δανείων και των καταναλωτικών δανείων. Και τη στιγμή κατά την οποία θέλουμε να αποκαταστήσουμε την ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν θα πρέπει να έχουμε δύο διαφορετικές νομοθεσίες. Θα πρέπει να έχουμε μια σωστή νομοθεσία στοχευμένη και τρίτον θα πρέπει οι κανόνες που αφορούν τα καταναλωτικά δάνεια να μην ε, εμπνέονται πάρα πολύ από την ε, πρακτική η οποία ακολουθείται για τα ενυπόθηκα δάνεια που ε, δεν έχουν ε, ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αρμόνιση πραγματική και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των στοιχείων τα οποία αναφέρουμε. Όταν μιλάμε για σφαιρικό ε, ευρωπαϊκό ε, τόκο ή ποσοστό να μιλούμε για συγκρίσιμα ποσοστά, για ποσά, διαφορετικά θα υπάρχει μεγάλη σύγκριση και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μη συγκρίσιμα μεγέθη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά την ψηφοφορία. Έχω την Περβόνς, τον Σλοβέρι, τον Ήτρα και βεβαίως θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Και μετά θα έχουμε και την έκθεση του κυρίου Μπάλτς για τον αθλητισμό. Σας υπενθυμίζω λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η διάταξη. Λοιπόν, ελπίζω ότι κάποιος θα μου δώσει τον κατάλογο των ε, ψηφοφοριών για να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ε, ας με σώσει η γραμματεία λοιπόν. Κατάλογος. Παρακαλώ. Είστε έτοιμοι. Έχουν ήδη διανεμηθεί σε όλες τις ομάδες οι κατάλληλοι ψηφοφορίες. Κανένας δεν θέλει να καθυστερήσουμε περαιτέρω. Αν είστε έτοιμοι και έχετε τις κάρτες σας, παρακαλώ. Ελέγξτε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Αρχίζει η ψηφοφορία, κάνουμε τεστ. Δοκιμή για να δούμε αν όλα δουλεύουν σωστά. Παρακαλώ. Τεστ. Okay. Okay. Right. Okay. So, uh, Λοιπόν, η πρώτη έκθεση, Λουτβίξεν, παράγραφος 1. Συμβαστική τροπολογία Α, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στην δεύτερη παράγραφο, συμβαστική τροπολογία Β, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Σ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η... Ψηφίζεται... Όχι. Όχι, δεν καταπίπτει η 7. Άρα την ψηφίζουμε. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το πρωτότυπο κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο έτσι όπως τροπολογήθηκε. Υπέρ. Θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ψήφισαν 40-36 προς 3 και μία αποχή. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα του 6802 εγκρίνεται. Αργότερα μπορούμε να ψηφίσουμε on block μόνο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ψηφοφορία, ε, τροπολογία α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτη συμβαστική τροπολογία εγκρίνεται. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορώ να ψηφίσω ο μπλοκ όλες τις συμβαστικές τροπολογίες ως το τέλος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Και τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Τώρα περνούμε στο σημείο 13, την έκθεση της κυρίας Οκονή, τυχερά παιχνίδια για απευθεία σύνδεση στην εσωτερική αγορά. Συμβαστική τροπολογία Α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογίας 13 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι έλλειξη ψηφοφορία. Καταπίπτει. Αποτέλεσμα ψηφοφορίας 20 προς 20. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο από την αίθουσα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το δεχθώ. Αυτό πρέπει να το αναγγείλετε πριν από το να μας το πείτε πριν την αγγελία του ψήφου. Εν πάση περιπτώσει καταπίπτει. Τροπολογία 31. Ε, Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία C. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. D. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι, έληξε ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συμβαστική ψηφοφορία εα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45. Υπέρ, κατά. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, επαλήθευση 45. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. 20 προς 20, καταπίπτει. Σέρπα, τι γίνεται. Ήσουν υπέρ. 22 προς 20 τότε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. G. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. H. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 42 η τελευταία τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πρέπει να ψηφίσουμε το κείμενο τώρα έτσι όπως τροπολογήθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έληξη ψηφοφορία. 38 υπέρ και 2 αποχές. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στην συνάδελφο Σοφή και πάλι. Όσοι θέλουν να αποχωρήσω από την αίθουσα, με ησυχία παρακαλώ, γιατί συνεχίζεται η συζήτηση. Σας δίνω δύο λεπτά για να βγείτε από την αίθουσα.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 Come on, get out, quick. Stop chatting. I think they've had long enough now, don't you? Okay, if we could have, we could have quiet. Λοιπόν, αν έχει την καλοσύνη, ησυχία, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ακούσει και τον εαυτό του που μιλάει. Επανερχόμεθα τώρα στη συνέχιση της συζήτησης για τις ε, υποθήκες ε, και ε, έχουμε λοιπόν άλλους τρεις που έχουν ζητήσει το λόγο και μετά τον εισηγητή. Η Πρεβόνς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα ενυπόθηκα δάνεια. Πρέπει να πω ότι βρίσκεται στα κάτω-κάτω σιρτάρ για τις Κομισιόν και πού και πού επανέρχεται. Υπάρχει όμως μια αντίφαση. Απ' την άλλη, απ' τη μία, όλοι θέλουν ε, να υπάρξει καλύτερη πολιτική σε θέματα ενυποθήκων δανείων, ώστε να μπορέσει η οικονομία να πάρει μπρος. Απ' την άλλη, κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει ότι η διαχείριση του συνόλου των ακινήτων είναι αυτή που οδήγησε και στην κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το θέμα αυτό. Δεδομένου ότι το θέμα αυτό των ε, ενυπόθηκων δανείων είναι πάρα πολύ. Γιατί όταν μας λέει κάποιος ότι 14 μέρες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για ένα τραπεζίτη, πιστεύω ότι ακολουθείται ένα ε, επιχείρημα το οποίο δεν νόμιζα ότι θα μπορούσα να το ακούσω το 2011. Τώρα, σε σχέση με τις προτάσεις του εισηγητή, πρέπει να αναγνωρίσω ότι δεν μπήκα στη λεπτομέρεια όσον αφορά όλε τι τροπολογίε που προτείνει. Γιατί τώρα αρχίζει η συζήτηση. Απλώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του σε δύο θέματα. Επέμεινε πολύ στο θέμα τη ε, οικονομικής παιδείας και ενημέρωση. Πολύ σημαντικό και σωστά το ανέφερε, αλλά για μένα η απόλυτη συμμετρία αυτή τη υποχρέωση είναι η υποχρέωση να παρέχονται οι σωστέ συμβουλέ. Pour l'offre de crédit hypothécaire d'être assortie, comme nous l'avons fait dans la MIF et comme nous devons le faire dorénavant dans toutes les offres de services financiers,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 pero que son referencias que sin duda alguna tienen un valor indicativo y lo que estamos planteando es sí, que existan como referencias y además en esto seguimos las recomendaciones. Και ακολουθούμε την σύσταση του Συμβουλίου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, διότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε συνεκτική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τώρα, για θέματα αμοιβών για τις διάφορες επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε σύγκρουση συμφερόντων. Όταν κάποιος παρέχει μια συμβουλή, το κάνει προς όφελος του πελάτη, του καταναλωτή και όχι για να μπορέσει για εμπορικούς λόγους να αποκομίσει κάποιο όφελος. Τώρα, η αξιολόγηση της ικανότητας πληρωμής. Επίσης δεν θα πρέπει να γίνει αντικείμενο εμπορίας. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα στοιχεία να αξιολογηθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Και το θέμα της ε, διαφήμισης είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την, Ευρωπαϊκή την ε, Επιτροπή εσωτερικής αγοράς. Διότι τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις μονίμως διαφημίζουν τα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα, τις τράπεζες, αυτούς που, που δίνουν τα δάνεια. Επίσης, το θέμα της δημοσιονομικής ποικιλότητα είναι σημαντικό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενοποίηση παντού. Θα πρέπει να θεωρηθεί η ποικιλομορφία ως ένα στοιχείο θετικό. De, de las hipotecas y favorece la inclusión en la medida que puede. El objetivo fundamental de un mercado desarrollado en el ámbito hipotecario es diseñar los productos atendiendo las necesidades de los consumidores y de los distintos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 in sport. And I can give apologies for Ramon Tremosa, who had to go to get his flight, and so he's not here as a shadow. But I'm sure we'll listen. Burkhard. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will es ja bewusst jetzt etwas knapper machen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Nach Can you be quiet if you're leaving, please?